Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, να αρχίσουμε. Έχω ανακοινώσει. Περίμενα να έρθουν οι συγητές. Βλέπω έναν άλλα. Ανακοινώσει θέλαμε να αρχίσουμε 9 παρατέταρτο, γιατί είναι πολύ βαριά η μερίσια διάταξη. Καθίστε παρακαλώ να σας κάνω τις ανακοινώσεις. Πρώτα έγκριση της ημερήσιας διάταξης φυσικά. Λοιπόν, για την ημερήσια διάταξη αυτή καθ' αυτή προτείνουμε τις εξής αλλαγές στο σημείο 7 για την κατάσταση στη Ρουμανία. Μετά από αίτημα της Ολομέλειας στις 8 Ιουνίου και της διάσκεψης των Προέδρων στις 11 Ιουνίου θα αρχίσει στις 3 αντί στις 11.30, το 8 στις 4 αντί στις 5 και τα 9 και 10 που είναι κοινή συζήτηση για την Ευρωπαϊκή η ε, Υπηρεσία Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα αρχίσει στις 11 αντί για τις 3. Με αυτές τις αλλαγές, αν δεν διαφωνείτε, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε. Η διερμηνία είναι στις εξής ε, ε, γλώσσες, όλες εκτός από δανικά, λετονικά, κροατικά και ιρλανδικά, ιδελικά. Σε 11 ψηφίζουμε, παρακαλείστε να έχετε έτοιμες τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Νομίζω ότι περιμένουμε συγγητή τώρα, συνεισηγητή, συνεισηγήτρια καλύτερα. Ε, μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν με το πρώτο βασικό θέμα, η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ε, συνολική, ολιστική, όπως λέγεται, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετανάστευση. Είναι πολύ σημαντική έκθεση και ενδιαφέροντες ομιλητές έχουμε για να δούμε όλα τα στοιχεία αυτής της έκθεσης. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, θέλω να εξηγήσω ότι ε, ποια είναι η πιο πρόσφατη κατάσταση ε, της έκθεσης, αντιμετώπιση των διακινητών ε, της Εκμετάλλευση των παράτυπων μεταναστών ε, και θα συζητήσουμε για την νόμιμη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων, τη θεώρηση διαβατηρίων, Frontex και το ρόλο του και άλλους οργανισμούς. Είναι έκθεση δίας πρωτοβουλίας. Βέβαια με την επιφύλαξη ότι σήμερα συνεδριάζει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρα και πάρα πολύ σχετικά. Καλωσορίσουμε τους προσκεκλισμένους μας, τον Δ. Γιώφτσοφ, πρώην Υπουργό Σωτερικών της Βουλγαρίας και ε, πρώην Διευθυντή της ε, Κρατικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας και το Wolfgang Ερ, που μόλις ευέστρεψε, που είναι δημοσιογράφος στη Zeit, εβδομαδιαία γερμανική εφημερίδα. Ε, θα συζητήσουμε για τέτοια θέματα, τράφικινγκ, ε, διακίνησης κτλ. Για το δεύτερο θέμα, πώς θα ε, προτείνουμε νόμιμους διάβλους για την οικονομική μετανάστευση. Έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων και τον καθηγητή Βαν Μάρτιν από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας για τη διαχείριση των συνόρων και την ε, θεώρηση διαβατηρίων και το ρόλο του Frontox και άλλων σχετικών οργανισμών έχουμε τον καθηγητή Steve Pierce του Πανεπιστημίου του Essex και την εξοχότητα του κύριο Ρομπέρτο Μπαλσαρέτη που είναι επικεφαλής της αποστολής της Ελβετίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας μιλήσει για την ελβετική ανθρωπιστική θεώρηση διαβατηρίων που ενδιαφέρει και τους συναδέλφους. Λοιπόν, θα δώσω πρώτα το λόγο τις ε, δύο συνεισηγήτρες. Βλέπω κατεύθυνση και η κυρία Σισίλ Κέγγε. Ε, λοιπόν, πρώτα οι συνεισηγήτρες, η Ρομπέρτα Μετσόλα και μετά η Σισίλ Κέγγε. Ρομπέρτα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Κλόντ, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους εξέχοντες ομιλητές μας που βρήκαν το χρόνο να έρθουν εδώ σήμερα. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Να δούμε τι θα κάνουμε για να ε, καταπολεμήσουμε τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών που ε, εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και ε, ε, τους ανθρώπους. Συζητούν σήμερα οι ηγέτες το θέμα αυτό και άρχισε αυτή την εβδομάδα και επιστολή UN, unaf 4 Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά τα δίκτυα του κακού όπου και να δρούν εντός και εκτός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική συνεργασία για επιβολή του νόμου και δίωξη. Ε, η διακίνηση ε, ανθρώπων και έχω συναντήσει πάρα πολλού εμπειρογνώμενου του τελευταίου μήνε, συχνά οδηγεί σε σεξουαλική εκμετάλλευση, εργατική εκμετάλλευση και ε, αναγκαστική επαιτία. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Χρειάζεται να ενισχυθούν οι δυνατότητε και οι επιχειρησιακέ δυνατότητε τη Europol συνδέονται τα δίκτυα αυτά με άλλες μαφίες και αυτό μας ανησυχεί. Τα δίκτυα αυτά, ξέρουμε, σπάνια δραστηριοποιούνται σε ένα κλάδο της εγκληματικής τους επιχείρησης. Έχουν κοινέ πληροφορίες, τις οποίες και διασταυρώνουν ε, ε, και εμείς πρέπει το ίδιο να κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη φάση μιας στρατιωτικής επιχείρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα βήμα. Οποιαδήποτε όμως επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα διακινδυνεύονται ποτέ οι ζωές των ε, προσφύγων και η αρχή της μη επαναπροώθησης θα πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστή. Πλην όμως, και αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό δεν θα πρέπει να ε, είναι βασισμένο στην ομοφωνία. Υπάρχουν κράτη-μέλη που θα πρέπει ε, να συμφωνούν για συγκεκριμένα μέτρα και ε, να μοιράζονται την αλληλεγγύη, να δίνουν ευκαιρία σε εκείνους που χρειάζονται προστασία, να τους δίνεται μια ελπίδα για το μέλλον χωρίς να χρειάζεται να πέφτουν στα νύχια αδίστακτων εγκληματιών. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι αυτοί οι άνθρωποι στην εκμετάλλευση γιατί ε, υπάρχει απειλή της σύλληψης και της απέλασης, άρα τους εκθέτουν σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να κυρώσει όλες τις συμβάσεις του Διεθνούς ε, ε, Οργανισμού Εργασίας για να προστατεύονται οι άνθρωποι αυτοί και να διώκονται όσοι τους εκμεταλλεύονται παντού και να μην υπάρχουν συστήματα που να ευνοούν τη μη αποκάλυψη, τη μη καταγγελία. Ε, δηλαδή, εδώ καλούνται και η κοινωνία των πολιτών και τα συνδικάτα, όχι μόνο οι ιδιοκτικέ αρχέ να δράσουν. Σε ό,τι αφορά του νόμιμους διάβλου, θα πρέπει να ξεφύγουμε από την Ευρώπη φρούριο και να δούμε ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε, όπω η λεγόμενη γαλάσια κάρτα στην Ένωση, για να ε, μετωπίσει τι ελλείψει. Αλλά να δούμε πού είναι και οι αδυναμίε και να καταλάβουμε ότι σε ένα μόνο κράτος συγκεντρώνεται η συντριπτική πλειονότητα όσων κατέχουν γαλάζια κάρτα. Δεν είναι λύση η ε, Ευρώπη φρούριο, αλλά ούτε είναι λύση να εγκαταλείψουμε τους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων. Δεν μπορεί να είναι ε, όμως η προστασία των συνόρων εις βάρος της ανθρωπιστικής μας υποχρεώσης να σώζουμε ζωές. Θα πρέπει ε, να δοθεί απαραίτητη σημασία και οι πόροι στους φορείς που το χρειάζονται. Ελπίζω η συνεισφορά σε σήμερα των εμπειρογνωμών να μας βοηθήσει και τη Σεσίλ και εμένα. Ευχαριστώ. Επόμενη συνεισηγήτρια, κυρία Σεσίλ Αγγέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση γίνεται την παραμονή μιας πολύ σημαντικής ε, συνάντησης από την οποία θα μπορούσε ίσως να προκύψει μια αλλαγή της προσέγγισης της Ευρώπης ε, στη μεταναστευτική ε, ροή ή μια συνέχιση ε, που θα αγνοεί τις ανθρώπινες ζωές. Μετά από τα πρόσφατα γεγονότα στη Μεσόγειο, φαίνεται ότι είχαμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει από πλευρά Ευρώπη. Σε αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ε, ανέθεσε περαιτέρω πόρου για την επιχείρηση Τρίτων και Ποσειδών και το γεγονό ότι ε, υπήρχε ένα πρώτο σχέδιο για του μετανάστε, ήταν ένα πρώτο ε, σχέδιο προ τη σωστή κατεύθυνση για μια κοινή και αλληλέγγυα μεταναστευτική πολιτική. Και επιτέλου μια καλή απάντηση από σε όσα είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν μια συμφωνία η οποία φαινόταν εύκολη, που ε, φαίνεται όμω όσο περνούν οι ώρε ότι χάνει την ουσία τη. Υπάρχουν κάποιε προτάσει οι οποίε θέλουν να αντισταθμίσουν τα αιτήματα υποδοχή ε, με την ασφάλεια των χωρών υποδοχή. Και φαίνεται η συζήτηση ότι θέλει να μετατοπιστεί από την ελληνική ε, με, σε καταπιαστικά μέτρα. Η Απέλπιδες προσπάθειες όμως των ανθρώπων που προσπαθούν να διαφύγουν από συγκρούσεις, από ένδια και από διώξεις ή απλώς ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον ε, δεν είναι απλώς ε, να ενισχύσουμε τα σύνορά μας, ούτε να έχουμε στρατιωτική ε, παρουσία στα σύνορα. Αυτές οι δράσεις απλώς και μόνο πιέζουν τους μετανάστες να κινηθούν σε πιο επικίνδυνες οδούς ή να εμπιστευτούν τη ζωή τους στα χέρια πιο επικίνδυνων διακινητών. Η καταπολέμηση λοιπόν του φαινομένου είναι ευθύνη μας και θα πρέπει να διαχειριστούμε τι αναστευτικέ ροέ των ανθρώπων που φτάνουν προ την Ευρώπη και να ε, δούμε τι γίνεται. Διότι το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει πλέον κατεπήγοντα χαρακτήρα, είναι διαρθρωτικό πρόβλημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για τα επόμενα χρόνια. Ε, διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν πολύ επιζήμιο πρόβλημα εάν δεν επιτεθούμε στα αίτια της διακίνησης. Η κατάσταση από τις χώρες τις οποίες διαφεύγουν ε, αυτοί οι άνθρωποι ε, είναι πολύ συγκεκριμένη και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με πρόσφυγες και ανθρώπους που χρειάζονται διεθνή προστασία. Δεν θα πρέπει να κλείσουμε την νόμιμη μετανάστευση στην Ευρώπη για οικονομικούς λόγους. Θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες μας σε αυτούς τους ανθρώπους που αναζητούν προστασία, αλλά και σε ένα νέο εργατικό δυναμικό, σε μία ήπειρο η οποία γυράσκει συνεχώς και εξακολουθούν να μειώνονται οι γεννήσεις. Μόνο οι νέοι λοιπόν μετανάστες ε, που αφήκνονται θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν το ποσοστό ανάπτυξης ε, ε, που φθήνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που αναζητούν θέσεις εργασία, να λάβουμε υπόψη τις μεταναστευτικές ροές και να ευνοήσουμε και κάποια προγράμματα προσωρινής μετανάστευσης. Θα πρέπει επίσης να διευρύνουμε και να πλουστεύσουμε τη διαδικασία εισόδου και αδειών διαμονή. Ε, των αλλοδαπών και θα πρέπει να δίνεται η γαλάζια κάρτα και σε εργαζομένους που δεν είναι υψηλών προσόντων. Για να υπάρχει νόμιμη μετανάστευση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια θα πρέπει να υπάρχουν και μέτρα και φιλόδοξες πολιτικές οι οποίες καταρχάς θα πρέπει να προσπαθούν να βοηθήσουν την ένταξη των μεταναστών και κατά δεύτερον την ελεύθερη κυκλοφορία των προσφύγων. Ελπίζω ότι οι εμπειρογνώμονες που βρίσκονται εδώ σήμερα θα δώσουν κάποιες μακροπρόθεσμες προτάσεις και για την ε, ε, υπεύθυνη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων. Δυστυχώς τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων έχουν φέρει στην επιφάνεια πολιτικές καταπίεσης, ε, κλειστές πολιτικές, κλείσιμο των συνόρων και προστατευτικά φράγματα. Το τι γίνεται με τους ανθρώπους που ζητούν άσυλο, η πρόβλεψη συστημάτων υποδοχής και χώροι υποδοχής οι οποίοι είναι εντελώς ακατάλληλοι και άνθρωποι που ζουν σε δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση αυτούς τους ανθρώπους ε, ε, που έρχονται. Δεν χρειάζεται τέτοιε πολιτικέ η Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να έχουμε ε, μελλοντικές προτάσεις για, για τον οργανισμό διαχείριση. Αναφέρομαι στο Frontex. Θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει συγκεκριμένα μέτρα. Κατ' εμέ θα πρέπει να στηριχθούμε σε άλλα μέτρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι μετασταυτικέ ροέ που προέρχονται από τη Μεσόγειο και όχι να έχουμε κατά μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, μιλητές τώρα. Ο Δόκτωρ Γιόντσεφ. Έχει πάνω από 10 λεπτά έκαστος για να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω σήμερα και να συζητήσω με τόσο σημαντικά ζητήματα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα προσπαθήσω να συντομία να σας ε, παρουσιάσω την κατάσταση, πώς αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες στη Βουλγαρία, την κρίση στη Μεσόγειο και να κάνω κάποιες προτάσεις για τις μελλοντικές ε, λήψεις αποφάσεων. Μία από τις βασικές αιτίες ε, της κρίσης είναι φυσικά οι ένοπλες σειράξεις στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολεί το ότι βραχυπρόθεσμα δεν πρόκειται να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Ε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι σε 4, 5, 10 χρόνια θα έχουμε ε, πάυση ένοπλες σε ε, Το αντίθετο μπορεί να είναι βαθύτερη η κρίση και οι χώρες γύρω από τη Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αποσταθεροποιηθούν όχι όχι μόνο με το, λόγω του αυξανόμενου αριθμού των προσφύγων σε αυτήν την περιοχή, αλλά για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Ο αριθμός των προσφύγων και παρανόμων μεταναστών θα συνεχίσει να αυξάνεται στο άμεσο μέλλον και βλέπουμε ήδη ε, ξεκάθαρα την τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλοί δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην πατρίδα τους αυτό θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, οπότε σύντομα θα πρέπει να καταρτήσουμε και να εφαρμόσουμε μια πρόσφορη στρατηγική. Ε, πρόκειται για μεγάλη πρόκληση για τη δική μας την ασφάλεια. Οι απειλές και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κρίση. Πρώτα απ' όλα ε, ε, υπάρχει ανθρωπιστική κρίση όχι μόνο καταβλισμός αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις, ε, συγκρούσεις, εθνοτικές και θρησκευτικέ συγκρούσεις, παραδοσιακή βία και δυσλειτουργία του κοινωνικού συστήματος. Φυσικά υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους και τη δική μας, το δικό μας πολιτισμό, προβλήματα επικοινωνιακά, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα μας και δεν έχουν τα μέσα στη διάθεσή τους, ούτως ώστε να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ε, και βασίζονται σε πηγές πληροφόρησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, χαμηλή κοινωνική διαστρωμάτωση, δεν... είναι άποροι αυτοί οι άνθρωποι, χρειάζονται υποστήριξη ε, διαρκώς, δεν έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, οι περισσότεροι είναι θύματα, υποφέρουν, έρχονται στην Ευρώπη και προσδοκούν ότι κάποιος θα τους αποζημιώσει για την προσπάθεια που έκαναν και θα έχουν τα ίδια επίπεδα διαβίωσης ε, με αυτά που είχαν νωρίτερα. Και δεν θεωρούν ότι πρέπει να δαπανίσουν χρόνο ή ενέργεια για να το πετύχουν. Ε, έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων για να βρουν μια δουλειά ε, περιορισμός της ελεύθερης μετακίνησης αυτών των ανθρώπων και αυτό οδηγεί σε ριζοσπαστικές τάσεις και φωναμενταλισμό. Επόμενη διαφάνεια. Αυτό δημιουργεί ε, προκλήσεις ε, για διάφορα ζητήματα, πόροι, χρήματα, ε, υποδομή, εξοπλισμός, οι δεξιότητες αυτών που έρχονται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, νέες τεχνολογίες, πληροφορίες όχι μόνο για αυτούς που είναι στους καταβλισμούς και διέρχονται παράνομα τα σύνορα αλλά ακόμη και για τις γενικότερες τάσεις και τις διαδικασίες, ε, κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερες ε, προγνώσεις και φυσικά για να κερδίσουμε χρόνο. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα μέσα, νέες διαδικασίες, ε, όμως γι' αυτό χρειαζόμαστε χρόνο. Ποια είναι η κατάσταση στην Βουλγαρία. Βλέπετε το 2013 την κόκκινη γραμμή 2014 ε, είναι η κίτρινη και 2015 η μπλε γραμμή. Για δείτε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2013, τότε εφαρμόσαμε την ενεργό πολιτική διαφύλαξη των συνόρων ε, για να αρχιτήσουμε την τάση. Βλέπετε όμως τα αριθμητικά στοιχεία το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι στιγμής βλέπουμε αυξανόμενη τάση και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Η Βουλγαρία έμπρακτα απέδειξε ότι με αποτελεσματικότητα μπορεί να διαφυλάξει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να βρούμε μια λύση στην κρίση, εξετάζουμε διάφορα μέτρα ε, προδραστική ε, πολιτική στα σύνορα. Ε, Στείλαμε συνοριοφύλακες, αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, ώστε να χειριστούμε καλύτερα ε, τα προβλήματα, αυξήσαμε τον αριθμό των καταβλισμών, 30 περισσότερους καταβλισμούς, ε, μάλλον κέντρα υποδοχής, ε, χρησιμοποιούμε περισσότερους πόρους για να αυξηθούν τα μέσα διαβίωσης τους και κάνουμε κοινά προγράμματα με τον ΕΑΣΟ και ευχαριστούμε τον ΕΑΣΟ και τον Frontex για τη σημαντική υποστήριξη που μας έχουν δώσει και με την, τον ΟΗΕ. Επίσης έχουμε επιτύχει χάρη σε αυτές τις προσπάθειες ε, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε κοιήσεις ε, ε, πλέον για την ασφάλεια όχι μόνο για του δικού μα πολίτε, αλλά γενικότερα για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δημιουργούμε μια στρατηγική ενσωμάτωση και κάνουμε ε, σοβαρέ προσπάθειε. Ελπίζουμε να τελεσφορήσει η προσπάθειά μα, εντατικοποίηση τη ε, και τη συνεργασία με τι γειτονικέ χώρε και ε, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες μας βοηθούν πολύ. Θα ήθελα να σας δείξω μόνο το ποιο αποτέλεσμα είχε η πολιτική μας τα σύνορα με αυτά τα νέα μέτρα. Περιμένουμε μέχρι τα τέλη του έτους να έχουμε περίπου 21.000 παρανόμες εισόδους. Ε, αν δεν είχαμε εφαρμόσει αυτή την πολιτική θα είχαμε ξεπεράσει τις 67.000. Τι σημαίνει αυτό για τρία χρόνια Πρόκειται για το 1% περίπου του πληθυσμού της Βουλγαρίας, για 10 χρόνια 3%. Δηλαδή μια μειοψηφία που δεν θα έχει ενσωματωθεί στην κοινωνία. Μπορούμε να το διαχειριστούμε δύσκολα. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ε, πολλά μέσα, πολλές προσπάθειες είχε κάνει ε, η Βουλγαρία και έχει αναλάβει δυσανάλογα μεγάλους κινδύνους για να διαφυλάξει ε, τα σύνορά μας, όχι μόνο για την Βουλγαρία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε, Ελλάδα και Ιταλία. Ε, ευχαριστούμε τους Υπουργούς Εσωτερικών, διότι διαχειρίστηκαν αυτή την καταστροφή. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Προτού ε, περάσουμε στην κρίση στη Μεσόγειο, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε κάποια, σε κάποιες επικίνδυες ε, είναι ε, τοπικό το πρόβλημα και άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, μέσα επί τόπου για να λύσουμε το πρόβλημα. Όχι, αυτό είναι, δεν ισχύει γιατί είναι περίπλοκη η κατάσταση και μπορούμε, πρέπει να κινηθούμε διαπεριφερειακά και διεθνώς μπορεί κάποιο να πει «Α, ναι, έχουν προβλήματα και στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και μπορούμε να τους βοηθήσουμε». Αυτή είναι αλληλεγγύη. Όχι, δεν είναι σωστή η προσέγγιση. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα Όλοι μαζί πρέπει να το λύσουμε. Δεν πρέπει να μιλάμε για αλληλεγγύη, για ευθύνη πρέπει να μιλάμε. Εάν δεν συνεργαστούμε και δεν υλοποιήσουμε επιτυχή μέτρα, μετά από λίγα χρόνια θα έρθουμε αντιμέτωποι, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλα τα κράτη-μέλη που τώρα δεν εμπλέκονται, θα έρθουμε αντιμέτωποι με πολύ πιο επικίνδυνα προβλήματα. Ε, η επόμενη παρανόηση είναι ότι είναι βραχυπρόθεσμο το πρόβλημα. Όχι, είναι μακροπρόθεσμο και χρειάζεται στρατηγική για να επιλυθεί. Δεν μπορούμε επίση ε, να βλύνουμε το πρόβλημα κρατώντα ε, του ε, πρόσφυγε στα κράτη-μέλη τη πρώτη εισόδου. Όχι, αυτό πάλι είναι επιστημονική φαντασία. Για δύο-τρία χρόνια μπορεί να γίνει αυτό, Όμω ούτω ή άλλω θα φτάσουν στον τελικό του προορισμό. Δεν θέλουν να μείνουν στη Βουλγαρία, θέλουν να ε, ε, εποφελθούν από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πλουσίων χωρών. Μετά από δύο-τρία χρόνια θα έχουν την άδεια μόνιμης παραμονής στη Βουλγαρία και θα το πετύχουν ή θα έχουν ακόμη και την υπηκότητα. Εάν εξακολουθούμε να κοιτάμε προς τη λάθος κατεύθυνση και να καταδαπανούμε τους πόρους μας ε, με μη πρόσφορο τρόπο, ξέρετε, θα έχουμε σε λίγα χρόνια ένα πολύ δυσχερές πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, ε, άλλη ε, πλημελής εντύπωση είναι ότι ε, μπορούμε να τους ενσωματώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, αυτό δεν ισχύει, διότι δεν είναι μόνο το πολιτισμικό χάσμα. Υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν να αποκτήσουν δεξιότητες, δεν θέλουν να ενσωματωθούν και δεν θέλουν να αλλάξουν κάτι. Γι' αυτό και είναι δύσκολη η διαδικασία ενσωμάτωσής τους. Δεν μπορούμε επίσης να θεσπίσουμε μια διαδικασία και να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε όλο αυτό το σύστημα. Μην ξεχνάμε τις βασικές αξίες Ευρωπαϊκής Ενωσίου σε κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόσφυγας ε, θα παραμείνει σε μια ε, γειτονική χώρα, λένε κάποιοι, αν ε, αναβαθμιστεί το επίπεδο διαβίωσης στο κέντρο υποδοχής. Ακόμη και πεντάστερο ξενοδοχείο, τέτοιο, τέτοιο επίπεδο διαβίωσης ε, διαβίωση να έχουν στα κέντρα υποδοχής δεν πρόκειται να μείνουν εκεί πέρα. Ε, δεν είναι δε μόνο το πρόβλημα των προσφύγων. 53% των αιτήσεων έχουν απορριφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ε, πάνω από 50% των ανθρώπων δεν έχουν κανένα συμφέρον να δηλώσουν πρόσφυγες. Έχουμε πρόβλημα γενικότερα με τους παράνομους μετανάστες. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, κανείς δεν ξέρει. Πόσους μετανάστες μπορούμε να πάρουμε επιτέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα εκατομμύριο, πιθανό. 20 εκατομμύρια δεν νομίζω. Ε, και αυτό είναι η πραγματικότητα. Βάσει της Eurostat για το 2012 έχουμε 1,7 εκατομμύρια νέες ε, πολιτογραφίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ε, είχαμε 660.000 ε, παράνομους μετανάστες και αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Πρέπει λοιπόν να ε, υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε κοινέ πολιτικές, να έχουμε περισσότερους πόρους για το, τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, για θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Ε, τώρα, μετά τα πρόσφατα γεγονότα δεν έχουμε αντιδράσει αρκετά γρήγορα. Βέβαια, λήφθη η απόφαση και ε, έκανε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμω χρειαζόμαστε χρόνο για να εφαρμοστεί η νέα πολιτική. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρέπει να λύσουμε και το θέμα των θεωρήσεων, των μονίμων τίτλων διαμονής, ε, των πολιτογραφήσεων, ε, του ασύλου Χρειαζόμαστε για συγκεκριμένες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αποτελεσματικότερες ε, πολιτικές, ε, χρειαζόμαστε πληροφορίες, κυρίως για τις υπηρεσίες διαχείρισης των συνόρων και ταυτοποίηση των μεταναστών, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι και θα τελειώσω. χρειαζόμαστε μια κεντρική ε, ε, πολιτική και κεντρική υπηρεσία ε, ασύλου και μετανάστευσης, αποτελεσματική υπηρεσία πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα εκτελεστικό οργανισμό για τις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασφάλειας. Κάποιες βάσεις τώρα για την πολιτική ενσωμάτωση από ε, κέντρωση, αποτελεσματική επικοινωνία, ε, επαγγελματικές ε, δεξιότητες, κοινωνική ενσωμάτωση και ζητώ συγγνώμη που μίλησα πάρα πολύ και τα είπα τόσο γρήγορα. Thank you very much um, Ευχαριστώ πολύ. Πάντα χρήσιμο είναι να έχουμε τέτοιες διαφάνειες και δομημένες ομιλίες. Συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά έχουν ζητήσει πολλά μέλη το λόγο και ε, θα ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο που έχουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δέκα λεπτά προσπαθείτε να περιορίζετε. Ξέρω ότι όλοι θα υπερβείτε το χρόνο σας. Ξέρω ότι θα μπορούσατε να μιλάτε μια μία ώρα και παραπάνω. Είναι τεράστιο το θέμα. Ε, παρακαλώ, όσο γίνεται περιοριστείτε. Ο κύριος Μπάουερ, θα γνωρίζετε ότι είναι δημοσιογράφος που έκανε έρευνα συμμετείχε στις μεταναστευτικές ροές ο ίδιος προσωπικά στην πηγή και έχει ζήσει από τα μέσα το πρόβλημα. Δεν το είπα στην αρχική μου ε, τοποθέτηση. Έχετε το λόγο λοιπόν κύριε Μπάουρ. Προτιμώ να μιλήσω γερμανικά προς αποφυγή παρεξηγήσεων και νομικών όρων και επειδή μου είναι και πιο εύκολο. Προτιμώ τα γερμανικά. Um, Νομίζω έχει παρέλθει ο καιρός που με αστυνομικά και στρατιωτικά μέτρα μπορούσαμε να περικαρακώνουμε τα σύνορά μας πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο, να το χωνέψουμε και προσπαθούμε να τον ανακτήσουμε. Αλλά με μέτρα ασφαλείας ε, και μόνο δεν πρόκειται αυτό να γίνει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι απελπισμένοι, η απόγνωσή τους είναι τόσο ε, μεγάλη, είναι τεράστια. Από ό,τι και να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα εξωτερικά της σύνορα, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, η Βουλγαρία ίσως έχει άλλη αντιμετώπιση γιατί με ένα σχετικό μικρό τείχος μπορεί να προστατευτεί. Ενώ τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιχαρακώνονται ε, με αστυνομικά μέτρα. Ως ρεπόρτερ έχω πάει εγώ τακτικά στη Συρία και έχω ζήσει την απόγνωση των ανθρώπων αυτών. Θυμάμαι κάτι βράδια, κάτι νύχτες στο Χαλέπι που είχαμε πέντε μαχητικά στον αέρα και διάφορα ελικόπτερα τα οποία ταυτόχρονα βομβάρδιζαν από ε, όλες τις κάνες και τα κανόνια που είχαν. Ο κόσμος, και εμείς το ξεχνάμε συχνά, ε, ε, παίρνει αυτά τα επικίνδυνα σκάφη και σαπιοκάραβα διότι κινδυνεύει η ζωή τους πολύ περισσότερο αν παραμείνουν στη χώρα τους από τον πόλεμο. Πριν από ένα χρόνο μεταμφιαστήκαμε σε πρόσφυγες από τον Κάφκασο, πήγαμε στην Αίγυπτο για να δούμε η διεισόμαση και να ζήσουμε στο πετσί μας πώς οργανώνεται η φυγή τους και τι σημαίνει. Στο μεταξύ έχει γίνει βιομηχανία η διακίνηση ε, ε, ε, και σε διαστάσεις κανονικά. Εγώ πάντα μιλάω για ε, μια σκιώδη βιομηχανία μεταφορών. 10.000 ε, στην Αίγυπτο είναι και μόνο αυτοί που οργανώνουν την επιμελητεία. Ε, υπάρχουν σε κάθε γειτονιά πράκτορες, διακινητές. Εμάς ήταν ένας εμπόρος επίπλων, συγγνώμη. Και μάλιστα σε θεωρούν πελάτη, σου τηλεφωνούν κιόλα και σου λένε έχουν καλύτερες διασυνδέσεις και και πιο φτηνή και ε, φτάνει στη θάλασσα όπου γίνεσαι όμοιρος πολύ γρήγορα. Τι άλλο ζήσαμε. Όχι μόνο οι διακινητές ευνοούνται και συγχρηματοδοτούνται ε, από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέψτε μου ε, ε, αυτό το σχόλιο και η Μπαλτασίρ που είναι η Αιγυπτιακή μαφία του κοινού ποινικού δικαίου, είναι εγκληματίε και προσπαθούν από τους διακινητές να κλέψουν ε, τους ε, πρόσφυγες και έτσι έγινε, μας απήγαγαν για τέσσερις μέρες μια μαφία με γυναίκες, παιδιά, 30 άτομα συνολικά ήταν η ομάδα των προσφύγων και μας φυλάκισαν μέχρι να πληρώσουν διακινητές νομίζω 3.500 στη μαφία για να μας αφήσουν ελεύθερους να μας ξαναπάρουν οι διακινητές. Η Αίγυπτος, κατά την άποψή μου, αποσταθεροποιείται μαζικότατα από την κατάσταση αυτή και αυτού του είδους την πολιτική. Συνέχεια μας συνέλαβαν στα παράλια της Αιγύπτου. Πήγαμε στις πρώτες πάρκες στη δεύτερη, στις τρίτες, ε, αλλά μας έβαλαν σε μία νησίδα, άμμο νησίδα, ε, γιατί δεν ε, κράτησε το λόγο του ο τελευταίος διακινητής, όπου μας έπιασε η αστυνομία Αιγυπτιακή 60 άτομα. Το μικρότερο παιδί ήταν 5 ετών και η πιο ηλικιωμένη γυναίκα 69 από την ίδια ομάδα. Όλοι μαζί σε 35 τετραγωνικά μας έβαλαν σε ένα χώρο σε ένα διαβόητο σοφρονιστικό κατάστημα, μια φυλακή της Αιγύπτου και ε, στο, ε, στο πάτωμα ήταν μπετόν, τίποτα δεν είχαμε και ακούγαμε όλη νύχτα αυτούς που φώναζαν από τα βασανιστήρια. Έχω βγάλει πολλά διδάγματα από το ταξίδι αυτό. Ε, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν οι διακινητές χωρίς να διπλασιαστεί ο κίνδυνος για τη ζωή των προσφύγων. Θα το θεωρούσα μέγα λάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να καταπολεμήσει τους διακινητές. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εμπορεύονται όπλα ή ναρκωτικά, αλλά με ένα πάρα πολύ εύθραυστο αγαθό που είναι το εμπόρευμα που λέγεται άνθρωπος. Και αυτό το εμπόρευμα πολλές φορές ε, χάνεται ή ε, στραπατσάρεται εντό εισαγωγικών όταν προσπαθεί να καταπολεμήσει διακινητές. Πολλού από του πρόσφυγες που γνώρισα προσωπικά, στη συνέχεια έγιναν διακινητές οι ίδιοι για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν το υπόλοιπο ταξίδι του γιατί κάποια στιγμή του τελειώνουν τα χρήματα. Ε, οπότε γίνονται διακινητές. Μιλώ για την Αίγυπτο. Στη Λιβύη η κατάσταση είναι πολύ πιο έντονη, πολύ πιο οξία και πολύ πιο τραγική από ό,τι στην Αίγυπτο. Έκτοτε λοιπόν αναρωτιέμαι Αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση. Είναι χήμερα να το πιστεύουμε. Γιατί δεν νομιμοποιούμε αυτό που τώρα γίνεται παράνομα. Αναρωτιέμαι γιατί συζητάμε χρόνια ολόκληρα για τα προγράμματα διάσωσης στη θάλασσα, αν θα διευρυνθούν, αν θα περιοριστούν, αφού στη δεκαετία του 90 ήταν πολύ επιτυχές το μοντέλο που είχαμε. Και είχαμε πάλι στις πόρτες μας ε, μπροστά στην αυλή μας ένα τεράστιο πόλεμο στη Βοσνία και τότε δεν υπήρχαν διακινητές, ούτε πέθανε ο κόσμος στα σύνορα, διότι είχε πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάτε. Επιτρέπετε, στο βαθμό που μπορείτε να αποδείξετε ότι κατάγεστε από τη Βοσνία, και γιατί στη Γερμανία, σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης, ε, χρειαζόμαστε ένα-δύο ε, υψηλά αμοιβόμενου υπαλλήλου για να κοιτάνε μήνες ολόκληρους αν είναι ε, ε, επικίνδυνη ζωή στο χαλέπι και να το αξιολογούν. Εγώ σας εγγυώμαι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δεν χρειάζεται ένα περίπτωση να ελέγχουμε αν είναι επικίνδυνη και να προσφέρουμε μια γενναιόδορη προσφορά και πρόσκληση να έρθουν οι άνθρωποι εδώ. Το έχουν κάνει ήδη γείτονε της Συρίας. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται αλλά μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, όπως ε, έγινε με τη Βοσνία μετά τη λήξη του πολέμου, να επιστρέψουν. Ε, εκατοντάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μάλλον ε, ήρθαν από τη Βοσνία και τώρα έχουμε δέκα χιλιάδες. Και εντάχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Δεν υπήρξε ακροδεξιά ολίσθηση στην κοινωνία γιατί θεωρούσε ο κόσμος ότι απειλεί το. Αν κάναμε λοιπόν κάτι τέτοιο, αυτόματα η βιομηχανία των διακινητών θα κατέρεε από μόνη της. Αν αυξήσουμε την πίεση στους διακινητές, τι θα γίνει. Ναι, ακόμα πιο αδίστακτοι χαρακτήρες και τύποι θα μπουν σε αυτή την πίσνα. Αυτοί που γνώρισα εγώ, ε, σε κάποιο βαθμό είχαν ένα ε, υπόλοιπο, ένα κατάλοιπο ανθρωπιάς και θα φύγουν αυτοί γιατί θα τους, είναι υπερβολικά επικίνδυνη αυτή η δραστηριότητα και θα μπουν εγκληματικοί τύποι σε αυτή τη δραστηριότητα που ε, δεν θα νοιάζονται για την ανθρώπινη ζωή, θα νοιάζονται ακόμα λιγότερο από τους σημερινούς. Σε αντίθεση με τον προλαλήσαντα πρέπει να πω ότι οι πρόσφυγες που είδα εγώ ε, είναι πολύ μορφωμένοι. Μιλήσατε εσείς για ανθρώπους χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Δεν ισχύει αυτό. Αυτοί που ήταν μαζί μου ήταν η μεσαία τάξη της Συρίας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ειδική οικονομική ζώνη μόνοι μας. Επιχειρηματίες από τη Δαμασκό με 500 υπαλλήλου παλαιότερα. Ήταν πανεπιστημιακοί, ε, απόφοιτοι, μηχανικοί, έχουν πολλές γνώσεις, είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και μπορούμε να χρειαστούμε και να αξιοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί οι άνθρωποι ε, επιθυμούν ε, διακαώς να έρθουν, αλλά θα πρέπει να τους αφήσουμε να το επιθυμούν αυτό και στην Ευρώπη, με ένα πρόγραμμα ένταξης και ενσωμάτωσης στην Ευρώπη. Περί τίνος πρόκειται αυτή τη στιγμή λοιπόν. Αυτό που επήγει είναι να σώσουμε ανθρώπινε ζωές και όχι κάποιες γραφειοκρατικές ε, διατάξεις και μεγαλόστομες δηλώσεις. Ο κόσμος πνίγεται μπροστά στα μάτια μας. Πνίγεται και μεταξύ άλλων διότι τους αφήνουμε να πνίγονται. Έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνη. Όχι μόνο το καθεστώς του κυρίου Ασάτ και οι ταραχές στην Μέση Ανατολή. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Για τις ζωές που χάνονται στη Μεσόγειο δεν επιτρέπεται να παραμένουμε ακόμα θεατές. Μια ολόκληρη νέα γενιά σύρων οθείται στην παρανομία. Δεν επιτρέπεται να τους ρίχνουμε στα χέρια και στα νύχια των διακινητών. Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν και την Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω την τάση ότι μας κάνουν πιο τραχείς ως κοινωνία ε, μας αλλάζουν. Σε λίγα χρόνια θα είμαστε διαφορετικοί. Προσπαθώντας να προστατευτούμε, αυτοκαταστρεφόμαστε. Τουλάχιστον οι αξίες και οι αρχές για τις οποίες βρισκόμαστε εδώ. Θυμάμαι ένα συνταξιδιώτη που ήταν στη φυλακή στην Αλεξάνδρεια μαζί μου, Μοχάμε τον έλεγαν, 30 και κάτι ήταν, ήθελε να πάει στη Σουηδία, δεν τα κατάφερε τον συνέλαβαν μαζί μας, τον άφησαν ελεύθερο, το ξαναπροσπάθησε, όπως και όλοι οι άλλοι σχεδόν. Ε, ξαναπήγε σε αυτά τα σκάφη και πέρσι το Σεπτέμβριο πνίγηκε. Μαζί με άλλους 500, εκ των οποίων 100 παιδιά. Και ελπίζω ε, να κάνουμε όλοι ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε στο μέλλον να μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα. ήταν εξαιρετικό άνθρωπος. Γιατί να πάει να πνιγεί στη Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στα πλαίσια της ε, νόμιμης ε, οικονομικής μετανάστευσης ε, και έχουμε τον κύριο Λούκα Βιζεντίνη εδώ. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι συναντήθηκαν μαζί του για την νόμιμη οικονομική μετανάστευση πριν από κάποιες μέρες. Ε, χαίρομαι λοιπόν που σας παρουσιάζω τον Λούκα και ε, του δίνουμε το λόγο για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο και τους συνεισηγητές ε, που κάλεσε την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ε, για να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Πρόκειται για μια συνομοσπονδία η οποία εκπροσωπεί όλα τα πιο σημαντικά συνδικαλιστικά σωματεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη και στις ε, γείτονες χώρες. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την έκθεση ίδια πρωτοβουλία για την μετανάστευση. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδίω αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για την κατάλληλη στιγμή για να συνεργαστούμε και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατεπίγουσα κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Επίση, πρέπει να πω ότι ενθαρρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σα πιο συγκεκριμένο να έχει όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή προσέγγιση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματο. γιατί υπάρχουν διάφορες πτυχέ που πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλες αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν στην ανάλυση. Ελπίζουμε ότι σήμερα η ατζέντα τη μετανάστευση που θα παρουσιαστεί από τον πρόεδρο Γιούνκερ θα εγκριθεί χωρίς να αποδυναμωθεί το περιεχόμενο του θεματολογίου, διότι η ατμόσφαιρα και η κατάσταση είναι ανησυχητική βάση και των απόψεων κάποιων κρατών μελών, αλλά εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας. Εάν εγκριθεί το θεματολόγιο, υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά θέματα τα οποία επιτέλους θα συζητηθούν, αν όχι και θα επιληθούν. Τουλάχιστον θα συζητηθούν. Η διάσωση στη θάλασσα αφενός και ε, η ε, κατανομή, το μοίρασμα των, τον άσυλο αφετέρου. Έχουμε περίπου 40.000 ανθρώπους ε, ε, από τη Συρία και την Ερυθρέα ε, και το φαινόμενο είναι ασυχητικό. Αλλά τουλάχιστον για μας αυτό θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης θα θέλαμε στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή δυνατόν να υπάρχει μια πίεση για μεσοπρόθεσμη τουλάχιστον αναθεώρηση για την οδηγία για τις επιστροφές και τη διάσωση και αναζήτηση και επίσης μια αναθεώρηση του κανονισμού του Διβλίνου για να γίνεται καλύτερη κατανομή των ετούντων άσελο και να είναι πιο σταθερή και πιο καλά διαρθρωμένη μεσοπρόθεσμα. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια του ασύλου. Καταρχάς θα πρέπει να ανοίξουμε νόμιμους διάβλους ε, για τους αιτούντες άσυλου, για να υπάρχουν ε, ε, προγράμματα δράσης για ανθρωπιστική βοήθεια, να επιτρέπεται να έρχονται κάποιοι άνθρωποι κάθε χρόνο, ένας αριθμός ατόμων και να μην πλήττονται από τη διακίνηση. Επίσης να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κατεπίγουσες καταστάσεις και να μην δίνουμε ταυτόχρονα μια όθηση στην εγκληματικότητα και στην παρανομία. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν νόμιμοι διευλοί για να υπάρχει καθεστώς ασύλου και στις χώρες ε, διέλευσης και διαμονής δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά αχ με συγχωρείτε χτυπάει και το τηλέφωνο μου. Συγγνώμη. Τρίτη παρατήρηση, τι θα θέλαμε να, έχουμε, να δούμε στην εκθεσή σας, να ε, μπορέσουμε να επιτεχύνουμε τη διαδικασία αναγνώρισης και ε, χορήγηση καθεστώτο ασύλου και να μην έχουμε αυτέ τι καθυστερήσει που έχουμε σε πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, πρέπει να ε, ανοίξουμε το δρόμο για να διευκολύνουμε την ένταξη των ε, μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασία. Καταλαβαίνετε ότι για μας ως συνδικάτα είναι πολύ ευαίσθητο το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίση, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί λίγο καλύτερα την εφαρμογή του κανονισμού του Διβλίνου και του κανονισμού Σέγγεν για να μην έχουμε ε, φαινόμενα όπω όπως ε, το Ουγγρικό ε, τείχος εντό εισαγωγικών και επίσης ε, ε, να μην επιτρέπεται σε κάποια κράτη-μέλη να παρακάμψουν ή και να αγνοούν τελείως τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Επίσης θεωρούμε ότι η αναθεώρηση για τους πρόσφυγες μπορεί να βοηθήσει τους, τις χώρες σε θέματα ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής. Υπάρχουν κάποια πρόσφατα παραδείγματα γερμανικών πρωτοβουλειών που μας δείχνουν ότι αυτή είναι η κατάλληλη λύση. Ε, πολλών μερών σε περιφερειακή περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων αυτών των ανθρώπων ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τώρα την οικονομική μετανάστευση που σχετίζεται με το θέμα των προσφύγων αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα ξεχωριστό ζήτημα. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βασίσει την ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που συζητούμε σήμερα σε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις. Όλα τα στοιχεία τα οποία παρέχονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από ανεξάρτητους φορείς ε, και ερευνητικά Ινστιτούτα καταδεικνύουν ότι η συνεισφορά των μεταναστών ε, στα δημόσια έσοδα των κρατών μελών όσον αφορά τη φορολόγηση και τα δημόσια έσοδα είναι πολύ σημαντικότερη από αυτά τα οποία λαμβάνουν ως κοινωνικά επιδέωματα και υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι ότι οι μετανάστες ου μόνον συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης ε, έρχονται να πληρώσουν το δημογραφικό κενό και ε, κάνουν πιο βιώσιμα τα συστήματά μας. Η προπαγάνδα που ε, επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για τον τουρισμό κοινωνικών επιδομάτων των μεταναστών είναι βάσει αυτών των στοιχείων εντελώς αβάσιμη. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι κάθε μακροπρόθεσμος μετανάστης ε, που εργάζεται ε, καταβάλει ε, αντίστοιχα ποσά και για τον εαυτό του αλλά για να καλύψει και άλλους ανθρώπους και το αυτό ισχύει και για νόμιμα εργαζόμενους μετανάστες γι' αυτό σημαίνει και ότι χρειάζονται και ίση μεταχείριση. Η μη καταγεγραμμένη μετανάστευση, μην την αποκαλείτε παράνομη μετανάστευση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν απλώ χαρτιά αυτοί, δεν είναι παράνομοι μετανάστε. Πρέπει να αντιμετωπιστεί καταλήλω, όχι με ε, σπασμωδικέ κινήσει. Αν ένα άνθρωπο εργάζεται ε, με. Ε, παράτυπε διαδικασίε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Αντί να τον απελάσουμε, θα πρέπει να τον προστατεύουμε και ο εργοδότη είναι αυτό ο οποίο θα πρέπει να τιμωρηθεί στη θέση του. Ε, επομένως θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή τη οδηγίας για τις κυρώσεις ε, και θα πρέπει να υπάρχουν και ε, έλεγχοι σε διαμεθοριακό επίπεδο ίσως. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ε, παράτυπη μετανάστευση και για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν ε, ε, έγγραφα και χαρτιά. Εμείς πάντα πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί και αυτή η πτυχή και θεωρούμε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση ίδια Πρωτοβουλία του θα πρέπει να το κάνει αυτό. Αντί να έχουμε μια κυκλική διαδικασία και μια επιλεκτική διαδικασία που έχουμε, έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει, θα πρέπει να έχουμε κατάλληλη πολιτική ώστε να προσελκύσουμε όχι μόνο εργαζομένους υψηλών προσόντων και τα ταλέντα που χρειαζόμαστε, αλλά όλες τις μορφές των εργαζομένων, διότι όλοι είναι χρήσιμοι. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη γαλάζια κάρτα, κατά την άποψή μας, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, διότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με λογικό τρόπο τις μεταναστευτικές ροές, πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Θα πρέπει να έχουμε πρωτοβουλίε οι οποίες θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν διάφορους τομείς. Ε, Παραδείγματος χάρη υγεία, προσωπική φροντίδα, ο κλάδος των τροφίμων, της γεωργίας, του τουρισμού. Και αυτοί οι τομεί δεν χρειάζονται μόνο άτομα υψηλών προσόντων. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ίση μεταχείριση προ του μετανάστε αν θέλουμε να αποφύγουμε ε, ε καταπίεση και να υπάρχουν, υπάρχει πλήρης ένταξη. Θα πρέπει να λαμβάνουν αντίστοιχο μισθό ε, όπως και οι εργαζόμενοι της κάθε χώρας. Επίσης πρέπει να υπάρχει πλήρη ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίε και δικαιώματα για τους μετανάστες σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι οι νόμοι μετανάστες που εργάζονται στην αγορά εργασίας συνεισφέρουν με τη φορολογία και τις κοινωνικές τους εισφορές όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα δικαιοσύνης, είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί και τα οικονομικά μας συμφέροντα ως Ευρωπαίους. Επομένως, η άνηση μεταχείριση δημιουργεί ε, αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων, διότι οι νόμιμοι ε, σε σχέση με τους παράτυπους έχουν τελείως διαφορετικά συστήματα και επίσης είναι και θέμα των δημοσίων αρχών. Εάν καταβάλλονται λιγότερα για φορολογία και κοινωνικές εισφορές ε, λόγω της παράτυπης εργασίας, αυτό σημαίνει ότι θα είναι και εις βάρος του δημόσιου προπολογισμού και δεν θα είναι βιώσιμα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ε, της κάθε χώρας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως Συνομοσπονδία Συνδικάτων ζητάμε πλήρως ίση μεταχείριση και ένα καλύτερο ορισμό του του ακριβώς συνιστά ίση στα διάφορα νομικά μέσα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα για τη μετανάστευση. Αυτά τα μέσα θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα μέσω μια κατάλληλη οδηγία και εξακολουθούμε να ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει προ αυτή την κατεύθυνση οι οδηγίες αυτές που δεν έχουν σαφώς εγγεγραμμένες αυτές τις, ε, ε, τις αρχές κατά την άποψή μας θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Η μεταρρύθμιση του συστήματος Schengen και θεωρήσεων διαβατηρίων μπορεί να είναι μια καλή ιδέα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν διακρίσεις και άνηση μεταχείριση για τα ε, συμβάσεις εργασίας ε, και τα συνθήκες μετανάστευσης. Τέλος, ε, δύο λόγια για το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και κυρίως των συνδικαλιστικών σωματείων στην μετανάστευση η Συνομοσπονδία των ε, Συνδικάτων και τα διάφορα δίκτυα των συνδικάτων παρέχουν συνδρομή, υποστήριξη και υπηρεσίες ένταξης στους μετανάστες, όπως επίσης κάνουν και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς και ενδιαφερόμενοι πέραν ε, της ε, δραστηριότητάς μας ε, σε πλαίσια διαπραγμάτευσης και πίεσης, οι υπηρεσίες αυτές είναι θεμελιώδεις για να βοηθήσουν τους μετανάστες, αλλά για να βοηθήσουν και τις δημόσιες αρχές να συνδράμουν τους μετανάστες. Ο, ο, ρόλος μας αυτός, λοιπόν, ο επικουρικός, πρέπει να αναγνωριστεί τρόπον τεινά και θα θέλαμε να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναφερθεί στην έκθεσή του σε αυτές τις συγκεκριμένε δράσεις, τις οποίες υλοποιούν διάφοροι οργανισμοί επιτόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Luca. And now... πάρα πολύ. Και τώρα ο καθηγητής θα μιλήσω ισπανικά. Γιατί έχουμε και μετάφραση, ωραία. Στο κέντρο μας, ε, εδώ και χρόνια εργαζόμαστε σε θέματα νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Και υπάρχει και Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση. Έχουμε policy briefs για την νόμιμη μετανάστευση Θέλω να δώσω και να στείλω μερικά σαφή μηνύματα και αν θέλετε, τηλεγραφικά και αν θέλετε στις ερωτήσεις να επεκταθούμε. Πρώτον, όταν γίνεται λόγος για σωστούς κατάλληλους διάβλους για νόμιμη εργασιακή μετανάστευση. Είναι ε, διαβλή που απαντούν στις ανάγκες ε, των ευρωπαϊκών οικονομικών και της αγοράς. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που εμείς τις έχουμε αναλύσει για το τι ανάγκες ε, σε εργατικά χέρια υπάρχουν στην Ευρώπη. Και συμφωνούν οι πάντες ότι για λόγους ε, τόσο δημογραφικούς όσο και δυνατοτήτων, προσόντων, δεξιοτήτων θα χρειαστεί η Ευρώπη εκατομμύρια νομίμων μεταναστών τα επόμενα χρόνια. Πάνω από 20 εκατομμύρια που ανέφερε κάποιος προηγούμενος speaker, ομιλητής δηλαδή. Είναι σημαντικό αυτό για την ευρωπαϊκή ευημερία ε, το επόμενο διάστημα. Θα αφήσουμε αυτό σε άναρχη εξέλιξη ή θα το ρυθμίσουμε ε, σύμφωνα με τις ανάγκες αγοράς. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε επίπεδο κρατών μελών, διότι τα κράτη-μέλη κατά τις συνθήκες έχουν την αρμοδιότητα να ορίζουν ποσοστώσεις νόμιμης μετανάστευσης. Ε, ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί βρισκόμαστε σε ένα χώρο με ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Και όπως ήδη αποδεικνύεται από την αγορά εργασίας, όταν έχεις ενοποίηση προς τα μέσα και κατακαιρματισμό της πολιτικής προς τα έξω είναι τεράστια τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών μέσα στην Ευρώπη, δηλαδή να έχουμε Ευρωπαίους με ελεύθερη κυκλοφορία και πολίτες τρίτων κρατών που στερούνται αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα σε μια ολοκληρωμένη επικράτεια. Οπότε... Έχει απόλυτη σημασία κάθε φορά να προσεγγίζουμε από πλευράς αγοράς εργασίας αυτό το θέμα της ε, μετανάστευσης που οφείλει να ενοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι θέμα δημόσιας τάξης αυτό δηλαδή όσο συχνά αντιμετωπίζεται. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε την νόμιμη τώρα μετανάστευση. Πρώτο, πολύ σημαντικό, πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί έτσι ώστε να συνδεθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των διαμενόντων ε, με την μετανάστευση. Το ίδιο ισχύει και με τους επιχειρηματίες. Δεν γίνεται καμία διάκριση. Ούτε συνταγματικά μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ μετανάστευση και ελεύθερη κυκλοφορία. Μπορεί να υπάρξει ένα σύστημα πανευρωπαϊκό ενημέρωση για τι ανάγκε τη αγορά. Υπάρχει σε εμβρική φάση με το σύστημα «Γιούρες» Ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσίων Υπηρεσιών Εύρεση Εργασίας, αλλά αυτό θα ήταν το μοναδικό εργαλείο που θα μας επέτρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε ένα είδος εξετάσεων που να εξασφαλίζει ε, ότι δεν έρχονται μετανάστες να υποκαταστήσουν ε, εργατικό δυναμικό που διαθέτει η Ένωση. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Ω τμήμα τη νόμιμη πάντα πολιτική μετανάστευση θα πρέπει να βρούμε μηχανισμού και μέτρα που να διευκολύνουν την ένταξη των μη οικονομικών μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφυγε φυσικά και εκείνους που έρχονται για οικογενειακή επανένωση, του ξένου φοιτητέ που έρχονται να σπουδάσουν. Είναι τρει κατηγορίε που καλύπτουν το 80% των μεταναστών στην Ευρώπη. Η οικονομική μετανάστευση είναι μόλις 20%. Θα πρέπει να βρούμε μέτρα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την νόμιμη μετανάστευση είναι κατακαιρματισμένη. Είναι λίγες οι κατηγορίες υψηλών δεξιοτήτων και προσόντων, εποχιακοί εργαζόμενοι, Ε, διαφόρων κλάδων εργαζόμενοι που κάνουν ανταλλαγές ε, θα γίνεται μια προσπάθεια να μειωθεί ε, η ροή των νομίμων μεταναστών αντί να δούμε τι ανάγκες έχουμε. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τις μεταναστευτικές ροές δεν έχει αλλάξει αυτή την προσέγγιση και εξακολουθεί να είναι χωρίς πραγματικό μακροπρόθεσμο όραμα για το τι ρόλο μπορεί να παίξει η νόμιμη μετανάστευση στο σύνολο της ευρωπαϊκής εργασιακής αγοράς. Κατά την άποψή μου, αυτό που χρειάζεται είναι πρώτον μια συνολική θεώρηση, να έχουμε όλη την εικόνα για την νόμιμη μετανάστευση. Σήμερα τη θεωρούμεθα. Το 2001 υπήρξε μια πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία απέρριψαν τα κράτη-μέλη και μήπως να την ξαναβρούμε. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος στη μεταναστευτική πολιτική, η εργασιακή μετανάστευση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ε, ότι οι εργοδότες χρειάζονται ε, εργατικά χέρια και να τα εξασφαλίσουμε αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, ε, οικονομικών μεταναστών που διαμένουν μόνιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σήμερα και νόμιμα. Σήμερα μπορούν να διαβούν τα σύνορα ως μετακινούμενοι Ευρωπαίοι πολίτες ας πούμε, αλλά όχι ως εργαζόμενοι. Επίσης, θα πρέπει οι που έχουν οι Ευρωπαίοι ε, να ε, καλύπτουν και τους άλλους πολίτες. Ας πούμε, εγώ είμαι Ισπανός, πήγα στη London School of Economics. Το πτυχίο μου αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες. Αν ήμουν Βραζιλιάνος ή από κάποια άλλη χώρα, Μαροκινός, δεν θα το αναγνώριζαν. Επίσης, η πρόσβαση νόμιμη στην αγορά ε, εργασίας στην Ευρώπη. Θα αναφερθώ και στη συνέχεια σε αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός θεώρησης διαβατηρίων για αναζήτηση εργασίας ορισμένων κλάδων ή κατηγοριών εργαζομένων, με συγκεκριμένα ειδικά προσόντα. Ήδη στη Γερμανία γίνεται και λειτουργεί έτσι, γενικά καλά. Και από την άλλη θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα μοριοδότησης ή έκφρασης ενδιαφέροντος, όπως ε, προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα δεν είναι πρόσφορο ε, ούτε καλύπτει τις ανάγκες. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Η Ευρώπη με 7 χώρες γειτονίας έχει συμφωνίες ε, μετακίνησης και μεταξύ αυτών είναι και η νόμιμη μετανάστευση και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προτείνει τίποτα ως νόμιμο διάβολο. σε πολλές από αυτές τις χώρες υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι με προσόντα ή και χωρίς ειδικευμένοι και ανειδικευτοί που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από τις εταιρικέ σχέσεις και αυτό θα έδινε και περισσότερη αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εξωτερική δράση προς τις χώρες αυτές που σήμερα λείπει. Έχω 1,5 λεπτό να αναφερθώ στο σύστημα μοριοδότησης ή ε, Έκφραση ε, εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έχει γίνει μεγάλος λόγος για το αυστραλιανό μοντέλο. Ποιο είναι το σύστημα μοριοδότησης. Είναι για την επιλογή των μεταναστών με βάση κάποια ε, αντικειμενικά κριτήρια που συνδέονται κυρίως με την ηλικία, τις σπουδέ, το επάγγελμα όπου θέτουν ένα ορόσημο για να πάρει άδεια εργασίας. Αυτό υπάρχει στη Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Αυστραλία και κατά κάποιο τρόπο πιο πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Το μέγα πρόβλημα ποιο είναι. Οι παραδοσιακές χώρες, αν ε, προσέξετε, ο Καναδάς και η Αυστραλία είναι μεγάλες χώρες αραιοκατοικημένες. Προσοχή εδώ. Και ε, έχουν ε, ένα σύστημα που υποαξιοποιούν τους μετανάστες, οι οποίοι έρχουν ε, τα προσόντα για να περάσουν το όριο αυτό της μοριοδότησης και να μπουν στη χώρα να δουλέψουν, αλλά μετά δουλεύουν ως ταξιτζίδες. Ε, κατά την άποψή μου λοιπόν, το σύστημα αυτό των μορίων δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο αυτό, θα υπήρχε κίνδυνος να ενταθούν ορισμένα προβλήματα που ήδη σήμερα έχει η Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας για διάφορους λόγους. Πρώτον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αξιοποιούμε ήδη τα προσόντα και τις δεξιότητες που έχουν άνθρωποι ειδικευμένοι. Εγώ είμαι από μια χώρα του πάνω από 20% των πτυχιούχων είναι ανέργοι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα σύστημα γενικά ε, πολύ γενναιόδωρο στις περισσότερες χώρες κράτους πρόνοιας. Οι νόμιμοι μετανάστες που θα περνούσαν αυτό το σύστημα μόριων δεν θα είχαν την απαραίτητη πίεση ή έναυσμα για να μπουν στην αγορά εργασίας αφού θα είχαν τα κοινωνικά επιδόματα και θα κινδύνευε έτσι να αυξηθεί ο αριθμός των ε, ειδικευμένων και προσοντούχων ανέργων που ήδη υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα καλύτερα να δούμε ένα σύστημα που να προσανατολίζεται στη ζήτηση, δηλαδή να έχει συμβόλαιο ε, εργασίας το οποίο να σου δίνει το δικαίωμα εισόδου στη χώρα και όχι το αντίστροφο. Ε, να φέρνουμε μετανάστε και να μην αξιοποιούμε τα προσόντα. Σταματώ εδώ για να μην σα φάω άλλο χρόνο και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Professor Martin. Καθηγητή Μάρτιν, να σας ευχαριστούμε. Τώρα ο καθηγητής Steve Pierce, ξέρω ότι πολλοί παρακολουθούν τις εργασίες του για τη διαχείριση των συνόρων, για την πολιτική των θεωρήσεων. Ε, Ασχολήθηκε με το Frontex, αν δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή ακρόαση. Πάντοτε χαίρομαι. Έρχομαι εδώ και να σας μιλάω για αυτό το θέμα. Δύο είναι τα βασικά σημεία που θα με απασχολήσουν, διαχείριση των συνόρων και θεωρήσεις. Για τις θεωρήσεις, Το σύστημα του Σέγγεν για τις θεωρήσεις έχει σχεδιαστεί μεταξύ άλλων και για βραχυπρόθεσμη διαμονή και εκεί υπάρχει ένα στοιχείο που θα μπορούσε να τροποποιηθεί και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως έχει για να καλύπτει και τις ε, αιτήσει για ανθρωπιστικούς λόγους, ε, για πιέσεις ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για όσους χρειάζονται διεθνή προστασία. Φυσικά τα κριτήρια του Σέγγεν για τις παραδοσιακές θεωρήσεις Σέγγεν καλύπτουν ε, το στοιχείο ότι υπάρχει πρόθεση επιστροφής. Υπάρχουν και διάφορα άλλα κριτήρια που ενδεχομένως δεν πληρούν οι ετούντες, αλλά σίγουρα οι ετούντες άσυλο δεν ε, έχουν αυτή την πρόθεση της επιστροφής, γιατί αλλιώς δεν θα ζητούσε κανείς διεθνή προστασία. Ενδεχομένως μακροπρόθεσμα να υπάρχει αυτή η πρόθεση, αλλά κυρίως πολύ μετά τη λήξη της βραχυπρόθεσμης θεώρηση ΣΥΝΙΕΝ μπορεί να υπάρχει ε, το σχέδιο να επιστρέψει κανείς στην πατρίδα του. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην περίπτωση των αιτήσεων ασύλου. Παρ' όλα αυτά, ο κώδικα θεωρήσεων και η σύμβαση Σέγγεν νωρίτερα, που αντικαταστάθηκε από τον κώδικα, προβλέπουν μια διαφορετική θεώρηση. Μια θεώρηση περιορισμένη εδαφική ισχύω. Περί τίνος πρόκειται περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, δηλαδή σε, ένα, σε μία από τις χώρες Σέγγεν που την εκδίδει. Από τη σκοπιά του Ετούντα αυτό δεν συνιστά πρόβλημα διότι παρέχεται η προστασία από ε, το κράτος που έχει εκδώσει τη θεώρηση και άρα βάση του χάρτη του Σέγγεν φέρει και την ευθύνη και μπορεί ε, να λάβετε και την άδεια διαμονής και να μπορείτε να μετακινηθείτε στο χώρο Σέγγεν ή αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψετε. Ε, ενδεχομένως πάντως να ισχύσει και για άλλες χώρες. Αυτό υπάρχει στον κώδικα όπως σας είπα. Και τι λέει ο κώδικας για τις θεωρήσεις. Ότι είναι περιορισμένη η εδαφική ισχύ αυτής της θεώρησης και υπό εξαιρετικέ περιστάσει για ανθρωπιστικού λόγου ή για άλλου λόγου διεθνού δικαίου μπορεί να διευρυνθούν τα κριτήρια αυτό, νομίζω κατά τη γνώμη μου, καλύπτει τους ετούντες άσυλο που ζητούν τέτοια θεώρηση. Και βάσει της διατύπωσης ε, υπάρχει μια υποχρέωση έκδοσης όταν πληρούνται ε, τα κριτήρια. Shall be issued, λέει ο κώδικας. Θα εκδοθεί η θεώρηση. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια απόφαση που λέγεται Προσκάκη, που είχε ζητήσει, ε, είναι ένας Ιρανός που είχε ζητήσει μια κανονική παραδοσιακή θεώρηση Σέγγεν και είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή όταν κάποιος πληρεί τα κριτήρια, πρέπει ε, οι αρχές να εκδώσουν για τη βραχυπρόθεσμη διαμονή την θεώρηση. Ο κύριος Κουρσχάκη ήθελε να πάει στη Γερμανία να επισκεφτεί τον αδελφό του που ήδη ήταν, είχε καθώς πρόσφυγα εκεί και οι γερμανικές αρχές τον υποπτευόντουσαν. Ίσως ε, θέλει να μείνει, ίσως έχει τα ίδια προβλήματα με τον αδελφό του και θα ζητήσει καθώς πρόσφυγα, οπότε καλύτερα να του τη δώσουμε τη θεώρηση. Και αυτό πυροδοτεί μια άλλη σκέψη, δηλαδή ε, μπορεί να υπάρξει ακτικότερη χρήση αυτού του συστήματος και δυνάμει ε, του κειμένου πλαισίου ενδεχομένως να χρησιμοποιείται συχνότερα από κάποια κράτη-μέλη, διότι υπάρχει και μια σχετική μελέτη, τη λάβατε πριν από λίγους μήνες, και απαριθμούνται εκεί οι κράτη-μέλη που ε, έχουν εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων υπάρχει νομική υποχρέωση για να εκδώσουν τη θεώρηση. Φυσικά εξατάται από την άποψη, την ερμηνεία του κώδικα Εκεί ενδεχομένως κάποια κράτη-μέλη έχουν λεπτομερέστερη διατύπωση, ερμηνευτική δηλαδή του. Θα έπρεπε σε ένα ξεχωριστό νομοθέτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ε, κατευθυντήριε γραμμέ και με κάποια χρηματοδότηση να ε, δοθούν απαντήσει για αυτό το ζήτημα. Διότι υπάρχει και το ζήτημα τη επανεγκατάσταση που ελπίζουμε σήμερα να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λοιπόν, εκεί ανοίγεται αυτή η προοπτική υποβολής αίτησης να έρθει κάποιο ως ετούν άσυλο σε ένα κράτος μέλος και να χρησιμοποιηθεί αυτό ως ισχύον νομικό πλαίσιο ε, όπου ε, προκύβει αυτή η νομική υποχρέωση. Αυτά για τις θεωρήσεις. Θα τώρα θα περάσω στα θαλάσσια σύνορα για τη διαχείριση των συνόρων. Υπάρχει ένα διεθνές νομικό πλαίσιο. Ε, είναι πάγια αμφιλεγόμενο το ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης της Γενέβης για όσους συλλαμβάνονται στα ανοιχτά ή στα χωρικά ύδατα και αποφασίζεται η επιστροφή τους. Τέλος πάντων δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση στην Ευρώπη διότι έχουμε την ε, νομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λέει ότι είναι εφαρμοστή η σύμβαση τουλάχιστον για τις συλλήψεις στα νυχτά και με το φαινόμενο της παρέκτασης ε, βλέπουμε ότι εάν ε, μπείτε στα χωρικά είδατα μιας χώρας ή εάν Ε, ασκείται έλεγχο επιτόπου μέσα στα πλαίσια των πολιτικών καταπολέμηση ε, των διακινητών. Αν τελικά εγκριθεί αυτό και γίνει στα χωρικά ιδιότητα της Λιβύης, Παραδείγματο χάρη, τότε έχετε την ευθύνη βάσει της απόφασης ε, του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν μπορείτε να στείλετε πίσω ανθρώπου σε χώρε που δεν είναι ασφαλεί και φέρετε και την ευθύνη για για μια περιορισμένη διαδικασία χορήγηση ασύλου, τόσο ώστε να μην επιστρέψουν σε επικίνδυνε χώρε. Δύο διαφορετικά νομικά πλαίσια λοιπόν στα οποία κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα δικά τη νομικά πλαίσια και έτσι εφαρμόζεται το ευρύτερο διεθνέ ε, ε, νομικό πλαίσιο για Το συντονισμό των θαλασσίων επιχειρήσεων του Frontex, κάτι που εγκρίθηκε πέρυσι, βλέπουμε ότι η θαλάσσια παρακολούθηση βάσει αυτού του πλαισίου έχει επεκταθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτή η νομοθεσία ενσωματώνει την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να επιστρέφουν κάποιες επικίνδυνες χώρες και πρέπει να τους δίνεται δυνατότητα να αποφαίνονται και βλέπουμε ότι υπάρχουν νομικές διατάξεις ερητέ στα πλαίσια των επιχειρήσεων θαλάσσιας παρακολούθηση. Υπάρχει βέβαια και το λεπτό ζήτημα, αν, όταν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο φέρει την ευθύνη για την εξέταση τη αίτηση ασύλου, διότι για τον κανονισμό του Δουβλίνου δεν είναι όσο εφόσον έχουμε βγει από τα χωρικά ύδατα των κρατών μέλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έρθει κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και ε, τους ε, συλληφθείς στα ανοιχτά και δηλώσει την πρόθεσή του να υποβάλει το αίτημα, τι γίνεται, θεωρείτε ότι έχει συλληφθεί ε, κοντά στα χωρικά είδατα της Μάλτας ή της Ιταλίας ή θα χρειαζότανε για όσους συλλαμβάνονται εκτός των χωρικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει ε, μία πρόνοια και για την, ε, τον επιμερισμό της ευθύνη και της ποσοστώσης μπορούμε να πούμε ότι όσοι συλλαμβάνονται εκτός των χωρικών υδάτων λοιπόν ε, εφαρμόζεται ένα, μία διαφορετική δέσμη κανόνων. Παραδείγματο χάρη η πρώτη χώρα εισόδου εκεί θα αποφασιστεί αν μπορεί να υποβληθεί ή όχι αίτηση. Λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα, ο συντονισμό των δράσεων από το Frontex. Υπάρχουν και αποστολέ των κρατών που δεν συντονίζει ο Frontex όμω, οπότε δεν θα ήταν ε, εν τη αυτή περιπτώσει εφαρμοστεί αυτό ο κανονισμό, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι παρεμφερή, διότι ο Συνοριακό Κώδικα Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί από τα κράτη-μέλη ίσως σε σημεία διέλευση να έχουν ε, επιχειρήσεις παρατήρησεις και τι γίνεται στην πράξη. Βλέπουμε ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και στα ανοιχτά αλλά και στα χωρικά ύδατα τρίτων χωρών διότι αυτό συνδέεται με το ρόλο του Frontex που πάλι επανασυνδέεται με τον συνοριακό κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Αυτά ακούσαμε στο προηγούμενο ε, Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και αυτή είναι και η άποψη του ε, Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Λοιπόν, ό,τι σχετίζεται με την εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζεται όχι μόνο σε ζήτημα ενωσιακού αλλά και διεθνούς δικαίου και άρα ενσωματώνει την ομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Δεν γίνεται να επιστρέψει κάποιο σε ασφαλή χώρα και πρέπει να του δώσετε τη δυνατότητα να σε εξηγήσουν γιατί δεν είναι ασφαλή η χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπουν οπωσδήποτε στην επικράτεια τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να πάνε, ξέρω εγώ, στο Μαρόκο, σε μια άλλη χώρα, εν πάση περιπτώσει, να, σε, να έχετε διμερή συμφωνία με τρίτε χώρε, ασφαλεί χώρε, ε, ο Μαρόκο, την Ισία, ούτω ώστε να ε, εξεταστεί ε, το αίτημά του σε ποια κατάσταση θα αντιμετωπίσουν αν επιστρέψουν. Αυτό είναι το ισχύον πλαίσιο. Θα μπορούσαμε με χρήσιμο τρόπο να το διευκρινίσουμε σχετικά με τα κριτήρια που αποφασίζουν ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο. Ε, από πλευρά του Frontex, ε, στο εγγύς μέλλον καλό θα ήταν να έχουμε νέε νομοθετικέ διατάξει. Ε, το ίδιο και για τις αρχές ε, των κρατών μελών, να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία στα πλαίσια του ελέγχου των συνόρων μετά από τις καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που έχουν γίνει για τις δράσεις των κρατών μελών και τέλος με τον συνοριακό κώδικα έχουμε νόμους, πρέπει να τους ξεκαθαρίσουμε απλώς και να είμαστε πιο να έχουμε μεγαλύτερη επιχειρησιακή ικανότητα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much, Professor. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Πίερς και ο τελευταίος ομιλητή μας είναι ο πρέσβης Ρομπέρτο Μπαλτζαρέτη ο οποίος πρέπει να εξηγήσει τη διαδικασία για την ε, θεώρηση ανθρωπιστικής ε, φύσεως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση και για την ε, πολύ σημαντική συζήτηση. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εγώ θα σταθώ σε μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή τον τρόπο με τον οποίο εφήρμοσε η Ελβετία τα τελευταία χρόνια αυτή τη θεώρηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο καθηγητής Πίερς έδωσε κάποια στοιχεία προηγουμένως. Εγώ θα επικεντρωθώ απλώς ε, στην πρακτική εφαρμογή της και λίγο στο ιστορικό. Καταρχάς, η ιδέα πήρε μορφή μετά από μια νομοθετική αλλαγή στην Ελβετία, η οποία επέτριψε στους ετούντες άσολο να υποβάλουν ε, αίτηση ασύλου στις ε, αντιπροσωπείες και στις πρεσβείες της Ελβετίας στο εξωτερικό. Ε, πρόκειται για μια νόμιμη διαδικασία λοιπόν με την αλλαγή της νομοθεσίας και λαμβάνει υπόψη της ε, κάποιες δύσκολες καταστάσεις και έτσι ο Υπουργός Πέθνος για τη Μετανάστευση στις 29 Σεπτεμβρίου του 2012 εξέδωσε μια εγκύκλιο η οποία επιτρέπει να Υπάρχει προστασία ε, με βάση τα στοιχεία της αίτησης ασύλου για ανθρώπους που διάκονται. Λόγω της κατάστασης στη Συρία, ένα χρόνο αργότερα, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2013, είχαμε ένα δεύτερο ε, μια δεύτερη οδηγία η οποία επιτρέπει να δεχόμαστε και μέλη της οικογένειας ε, του Σύρου ζητούντα άσυλο, ο οποίος ε, έχει λάβει αυτή την ειδική, ε, την ειδική θεώρηση ή έχει λάβει υπηκότητα στην ε, Ελβετία. Και έτσι λάβαμε υπόψη μα την κατάσταση στη Συρία και το τελευταίο διάστημα χίλια άτομα μπόρεσαν να έρθουν στην Ελβετία βάσει αυτής της ανθρωπιστικής θεώρησης. Η Ελβετία έχει δώσει θεώρηση σε 4.673 άτομα από τη Συρία και σε 200 άτομα τα οποία δεν είναι υπήκοοι Συρίας. Πώς έχει η, η διαδικασία. Πρόκειται για μια συνήθη διαδικασία που επιτρέπει στην αντιπροσωπεία, στην πρεσβεία που βρίσκεται στο εξωτερικό να εξετάσει τα αίτια τα οποία, για τα οποία υποβάλλει αίτηση ο συγκεκριμένος υποψήφιος. Αν θεωρήσει ότι δεν είναι ανθρωπιστική λόγη, απορρίπτεται η αίτηση. Αν θεωρήσει όμως ότι τα αίτια είναι ανθρωπιστικής φύσεως ή αν υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, το αίτημα διαβιβάζεται στις κεντρικές αρχές στην Ελβετία, οι οποίες αποφαίνονται για τα αίτια και από εκεί και πέρα επιτρέπουν την έκδοση αυτής της ειδική θεώρησης. Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία και επίσης υπάρχει και μια πιο ιδιαίτερη διαδικασία που αφορά την ιδιαίτερη περίπτωση της Συρίας και αποφασίστηκε ε, το Μάρτιο του 2015 από την κυβέρνησή μας που επιτρέπει στους ανθρώπους που πλήττονται από την ε, ε, Συριακή σύρεξη και ζουν στην Ελβετία να ζητήσουν από τις ομοσπονδιακές αρχές θεώρηση για τα μέλη της οικογένειας τους, δηλαδή τη σύζυγο, το σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα. Εάν κάποιος θέλει να έρθει λοιπόν ε, ε, στην Ελβετία μπορεί να έρθει να επανενωθεί με τα μέλη της οικογένειας, ε, με τον άνθρωπο ο οποίος έχει λάβει υπηκότητα στην Ελβετία. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία που επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να λάβουν αυτή την ειδική θεώρηση ο καθηγητής ε, Πίερ σας εξήγησε ότι επιτρέπεται η έκδοση ε, τέτοιων θεωρήσεων βάσει του κώδικα Σέγγεν. Εμείς ε, συζητήσαμε και με τις υπόλοιπες χώρες ε, το σύστημα Σέγγεν. Υπάρχει μια εθνική θεώρηση, μια θεώρηση τύπου Δέλτα, έτσι όπως λέει, αποκαλείται. Πρόκειται για τη θεώρηση η οποία θα πρέπει να δίνεται εξ αρχής σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι όπως είπε και ο καθηγητής Πίας, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην Ελβετία με αυτή την ανθρωπιστική διαφορετική θεώρηση και δεν ε, χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων όμως. Εμείς αποφασίσαμε ένα διαφορετικό σύστημα να δίνεται μια θεώρηση Σέγγεν, περιορισμένη σε δαφικής όμως ε, χρήσης που ισχύει μόνο για την Ελβετία και ισχύει για το κώδικα Σέγγεν για, τους δύο, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όταν δίνεται θεώρηση Σέγγεν αυτός ο οποίος λαμβάνει τη θεώρηση δίνει τα δακταλικά του αποτυπώματα και έτσι είναι πολύ εύκολο να γίνει μια αναζήτηση ε, για τις περιπτώσεις τις οποίες ε, ε, μπορεί στο μέλλον να υποβληθεί αίτηση ασύλου. Έτσι θα είναι ενταγμένος και καταχωρισμένος στο σύστημα. Και ο δεύτερος λόγος, αντίθετα με τις θεωρήσεις τύπου ΔΕΛΤΑ που δίνουν πρόσβαση σε όλο το χώρο Σέγγεν, αυτές οι θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικότητας δίνουν πρόσβαση μόνο Επομένω, στην Ελβετία. Επομένως είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε εμεί αυτή την, ε, στην περίπτωση γιατί ε, στις περισσότερες περιπτώσεις ε, σαφώς δεν πληρούνται ώρες οι προϋποθέσεις από τους ετούντε για να μπορούν να κυκλοφορούν στο χώρο Σέγγεν. Από το Μάιο του 2015 θα έχουμε αυτές τις ειδικέ ε, θεωρήσεις και καλέσαμε και άλλα ε, κράτη-μέλη του Σέγγεν ε, να μας πούν την άποψή τους για το θέμα αυτό. Εξετάσαμε την πρακτική εφαρμογή και εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ανάγκη προσαρμογής θα τις προσαρμόσουμε. Αλλά θα θέλαμε να σας πούμε ότι αυτή η πρακτική της Ελβετίας να δίνει αυτές τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις είναι μια λύση για να λαμβάνει υπόψη την κατεπίγουσα κατάσταση και τα ανθρωπιστικά προβλήματα που υπάρχουν και λαμβάνει υπόψη υπόψη της και τις νόμιμες διατάξεις. Αυτές οι συγκεκριμένες θεωρήσεις που είναι περιορισμένης ε, εδαφικότητας ε, έχουν ως προϋπόθεση να δίνονται δακτυλικά αποτυπώματα και σε καμία περίπτωση δεν θέτουν σε κίνδυνο το σύστημα Σέγγεν. Η Ελβετία είναι υπεύθυνη για πιθανό αίτημα ε, ασύλου το οποίο μπορεί να υποβληθεί μετά την άφηξη του εν λόγω ατόμου στην Ελβετία. Επειδή αναφερόμαστε στη ΣΕΓΕ, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να προσθέσω και κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό και να αλλάξω λίγο θέμα. Είναι προς το συμφέρον της Ελβετίας ε, να υποστηρίξει με αλληλεγγύη τις χώρες τις οποίες το καθεστώς ασύλου και υποδοχής ε, προσφύγων υπόκειται πολύ μεγάλες πιέσεις και αυτό μέσω του συστήματος του Δουβλίνου. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ασύλου, της ΕΑΣΟ και να ενισχύσουμε το σύστημα ασύλου στην Ευρώπη. Ε, συμμετέχουμε ατύπως ε, στις εργασίες αυτής της υπηρεσίας, παραδείγματο χάρη στην ομάδα για τη χώρα καταγωγής ε, και σε επιχειρησιακά ζητήματα. Το Μάρτιο του 2015 το κοινοβούλιο μας δέχτηκε τη συμφωνία ΕΑΣΟ την οποία συνάψαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του ασύλου για την Ελβετία και για τη συμμετοχή της Ελβετίας στις δραστηριότητες της ΕΑΣΟ. Ε, η συμφωνία θα κυρωθεί από τον Ιούλιο και από εκεί και πέρα ε, θα ε, ξεκινήσει να εσχέει και θα εκπνεύσει και η υποχρέωση για δημοψήφισμα. Δεν θα χρειαστεί λοιπόν δημοψήφισμα για την εγκρίνουμε. Το, η Ελβετία λοιπόν περιμένει απόφαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συμμετέχει και η Ελβετία σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much to, um, all... Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και την προσοχή που δείξατε. Θα ήθελα τώρα ίσω να δώσω το λόγο στις συνεισηγήτριες. Το λόγο, αλλά πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τους σκιώδης ε, Χέλγκα Στίβενς από το ECR. Δύο λεπτά έκαστος ε, παρακαλώ. Όλοι είναι στον κατάλογο το άλλως. Ακόμη και να μην θέλετε θα μιλήσετε όλοι και εσείς είστε. Και εσύ Τζούντιτ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα πολλές από τις τοποθετήσεις ακούσαμε για διακινητές, για διακίνηση ανθρώπων, για οικονομική μετανάστευση, πολλά θέματα αναφέρεται. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να σταθούμε. Και για την οικονομική μετανάστευση άκουσα ότι χρειάζονται προϋποθέσεις και όροι. Στην Ευρώπη ξέρουμε την οδηγία για τη γαλάζια κάρτα και νομίζω ότι είναι ένα καλό εργαλείο. Αλλά όταν συζητούμε για την οικονομική μετανάστευση και κοιτούμε τι γίνεται και με την οδηγία για τη γαλάζια κάρτα, πάντα πρέπει να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο. Υπάρχουν άνθρωποι με προσόντα, μορφωμένοι, ε, που ψάχνουν δουλειά, αλλά η γαλάζια κάρτα έχει μια πολύ βαριά διαδικασία για να χορηγηθεί. Ε, όταν θέλεις να ε, δώσεις εργασία σε έναν άνθρωπο με γαλάζια κάρτα, έχει υψηλότερο μισθό από τον κανονικό. Αλλά εσείς μιλάτε για νέους που ψάχνουν δουλειά ε, και είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου ή τεχνικών σχολών χωρίς να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κοιτάξουμε τα κριτήρια λοιπόν της γαλάζιας κάρτας πρέπει να τους πληρώνεις περισσότερο. Ποιος εργοδότης θα δώσει ευκαιρία σε τέτοιους ανθρώπους γνωρίζοντας ότι παίρνουν μια μισή φορά το μισθό του κανονικού υπαλλήλου. Ε, είναι άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία, μπορεί να έχουν ένα μορφωτικό επίπεδο και γνώσεις, αλλά πρέπει να τους προσλάβεις περισσότερο. Ενώ με λιγότερα χρήματα μπορείς να προσλάβεις κάποιον πολίτη της Ένωσης με εμπειρία κτλ. Δεν ξέρω, μήπω πρέπει να, να προσαρμοστεί αυτό το σύστημα της γαλάζιας κάρτας. Θέλω να σας, γνωρίσω, να σας ρωτήσω συγγνώμη, την άποψή σας. Για τους διακινητές συμφωνώ απολύτως με όλα αυτά που ακούσαμε. Ε, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Υπάρχουν όμως και άλλα υποκείμενα αίτια Άκουσα πολύ καλά αυτό που είπατε, ότι θέλουν να έρθουν πολλοί στην Ευρώπη ως οικονομικοί μετανάστες. Βεβαίως, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Αλλά ο κύριος Μάρτιν, ο καθηγητής, είπε ότι... Τι είπατε για την Ιταλία, όχι, κάπως Ότι υπάρχουν άνθρωποι πτυχιούχοι και το 20% είναι άνεργοι στη χώρα σας, στην Ισπανία. Στην Ισπανία, όχι στην Ιταλία. Τι γίνεται στις άλλες χώρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί πτυχιούχοι που είναι άνεργοι τελικά γιατί δεν βρίσκουν δουλειά σύμφωνοι με τα προσόντα τους. Και ταυτόχρονα μας λέτε να ανοίξουμε την αγορά εργασίας για ανθρώπους που έρχονται εκτός της Ευρώπης. Ε, θεωρητικά αυτό είναι καλή ιδέα, αλλά δεν φτάνει η δουλειά που έχουμε για τους ανθρώπους του δικού μας. Πώς να ανοίξουμε τις θύρες για τους εξωτερικούς με όλε τι καλές προθέσεις. Κοιτάξτε τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Κάντε μια βόλτα στις Βρυξέλλες να δείτε πώς οι νέοι άνεργοι είναι αργόσχολοι στο δρόμο. Και να έρθουν κι άλλοι. Αυτό είναι κάπως προβληματικό για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τους ομιλητές που έρχονται για πρώτη φορά θα ακούσετε σχόλια και ερωτήσεις. Παρακαλώ σημειώστε τις ερωτήσεις που απευθύνονται σε εσά για να απαντήσετε στο τέλος. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε όλα, σε κάποιο βασικά όταν τελειώσουν οι μιλητές. Η Σεσίλια Βίξτρομ από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές πολύ ενδιαφέρουσε παρουσιάσει σα για, το λαθρεμπό... για το εμπόριο ανθρώπων. Ναι, είναι ε, μια δουλειά που βασίζεται στην εκμετάλλευση των ανθρώπων οι οποίοι χρωστάνε για ολόκληρη τους τη ζωή και κινδυνεύουν. Ορισμένες φορές δεν έχουν όμως άλλη επιλογή αυτοί οι άνθρωποι και ανθίζει αυτή, αυτό το εμπόριο, θέλετε, διότι είναι ε, μονοπόλιο, δεν έχουν άλλη λύση αυτοί οι άνθρωποι. Επιστρέφω στα βασικά λοιπόν. Πώς γίνεται να έχουμε μια άλλη εναλλακτική λύση, νόμιμη και ασφαλή. Διότι οι περισσότεροι είναι προφανές θα επέλεγαν αυτή την εναλλακτική λύση. Αν υπήρχε, δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τους διακινητές σε καμία περίπτωση, αν δεν ε, παράσουμε μια τέτοια εναλλακτική λύση. Για την μετανάστευση, την πάνω μετανάστευση, πρέπει ουσιαστικά να συνδεθεί με το άσυλο, διότι υπάρχουν ε, διασυνδέσεις στην πράξη. Θα σας δώσω ε, ένα παράδειγμα. Ένα τρίτο των αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο κ. μας το είπε, προέρχονται από ανθρώπους από τα Δυτικά Βαλκάνια. Το ποσοστό απόρριψης αυτών των αιτήσεων ε, ανέρχεται περίπου στο 100%. Παρ' όλα αυτά όμως συγκαταλέγονται στα στατιστικά μας στοιχεία. Από το 53% απορρίπτεται. Δεν ε, επεξεργαζόμαστε αυτές τις αιτήσει. Πρόκειται για αιτούντες άσυλο, αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλουν δεν είναι άσυλο, είναι να βρουν δουλειά. Οπότε, ε, είναι τέτοιο το μέσο που παρέχουμε για την πρόσβαση ε, στην αγορά εργασίας που είναι ευκολότερο για αυτούς να ζητήσουν άσυλο παρά να μπουν στην περίπλοκη διαδικασία και τους περίπλοκους κανόνες για την νόμιμη μετανάστευση. Βλέπε οδηγία για εποχιακούς εργαζόμενους. Εάν υπάρχουν ελκυστικοί κανόνες για την νόμιμη μετανάστευση, ταυτόχρονα θα περιοριστεί ο αριθμός των μη στοιχειοθετημένων αιτήσεων εσύλου που απορρίπτονται. Θα λειτουργεί πιο καλύτερα το σύστημα και όσοι χρειάζονται την προστασία θα έχουν ένα ε, καλύτερο σύστημα. Ελεύθερη μετακίνηση τώρα. Είναι επίσης απαραίτητο σε αυτό το πλαίσιο να το εγγυηθούμε. Πρέπει να βλέπουμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα τα, τα πράγματα. Κανείς δεν σας δεν αναφέρθηκε σε αυτό με τον ε, γυράσκοντα πληθυσμό, με τις καταστροφικές δημογραφικέ τετάσει. Ε, θα χρειαστούμε ξένα χέρια στην αγορά εργασίας. Ακόμη και το Συμβούλιο το είπε στην ανακοίνωσή του. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως άλλως το έχει πει. Όμως ε, προσπαθούμε μόνο να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις ε, και δεν ασχολούμαστε με να προσελκύσουμε αυτούς που θα χρειαστούμε στο μέλλον. Θα έχουμε πελώρια προβλήματα. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο το σημερινό πρέπει κάτι να κάνουμε τώρα. Καθηγητή Πύρης δεν μπορείτε να επανέλθετε σε αυτό. Πολύ θα με ενδιέφερε να ακούσω την άποψή σας ε, τι δημογραφικέ τάσει που παρατηρούμε σήμερα, πώ ακριβώ θα τι χειριστούμε στα πλαίσια τη εντολή που έχουμε σήμερα. Ε, θα ζητούσα, λέει ο Πρόεδρος, ε, από τους ομιλητές ε, να απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα, διότι πρόκειται για πάγια ερωτήματα. Δεν θέλω δηλαδή να κάνετε καταληκτικές παρατηρήσεις, θέλω να απαντήσετε σε αυτά που σας ρωτάνε. Η Εύα Ζολή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Ε, διότι μοιράζονται την, ε, τις τεχνικές τους γνώσεις μαζί μας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάουρα που μοιράστηκε την εμπειρία του μαζί μας, μας εξήγησε τι, πώς, είναι, πώς είναι να ζει κανείς στο παιδί του την περιπέτεια του πρόσφυγα. Ε, τι έγινε στις 23 Ιουνίου με το ηλιοστάσιο στα ανοιχτά της Λιβύης. 2.800 πρόσφυγες ε, ε, βοηθήθηκαν από τους Ιταλούς συνοριοφύλακες, όμως έφτασαν και περιβολισμοί σε ένα από τα σκάφη, ένας πρόσφυγας πνίγηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ιταλία. Ξέρετε ότι εμείς οι πράσινοι είμαστε κατά της στρατιωτικοποίησης ε, του, του κυνηγιού αυτού κατά των διακινητών, διότι θεωρούμε ότι αυτό επιδεινώνει τη θέση των μεταναστών. Και δεν μπορώ παρά να ε, μνημονεύσω ε, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το 1942 η Ελβετία έκλεισε τα σύνορά της στους Εβραίους, διότι φοβόταν, δεν έχει να τους τρέψει. Φοβόταν ότι δεν έχει να τους δώσει δουλειά. και ότι θα εξευρωποιεί το, το, ο πληθυσμό της. Παρόμοια είναι η σημερινή κατάσταση για τους Σύρους. Δεν τους αφήνουμε να μπουν στις χώρες μας, τους απορρίπτουμε και εκείνοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Για θυμηθείτε, εμείς τότε δεν θα θέλαμε η Ελβετία να είχε βοηθήσει περισσότερο, να είχε αποτρέψει ένα μέρος της γενοκτονίας. Εύκολο είναι μετά να κλαίμε και να θρυνούμε. Είναι παρόμοια κατάσταση σήμερα. Θέλω να τους υποδεχόμαστε θερμότερα και για δημογραφικούς λόγους τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα το να έρθουν ε, μετανάστες με ε, ψηλή ειδίκευση είναι μια επένδυση για το μέλλον. Θα ήθελα να ε, ρωτήσουμε ε, να, επίσημα την Ιταλία τι έγινε με την έρευνα για αυτή την ανθρωποκτονία και να αποφύγουμε την στρατιωτικοποίηση ε, του ε, κυνηγιού κατά των διακινητών. Ευχαριστούμε, Εύα. Η Μάλιν Μπιόρκ τώρα για τη UNGL. Ευχαριστώ. Η ισχυρότητα μας η Μπάρμπαρα Σπινέλη δεν μπορούσε να έρθει, θα τα πω εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Ε, νομίζω ότι βλέπουμε διαφορετικές απόψεις και πολύ πιο διαφορετικές από τα... το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που διαβάσαμε χτες και προχτές. Τι βλέπω στα συμπεράσματα είναι λανθασμένο το εφαλτήριο και άρα καταλήγουμε και σε λανθασμένες λύσεις. Συμφωνώ με τους πράσινους, ε, δεν είναι μέρος της λύσης το να θα απλά και μόνο στους ε, διακινητές. Ε, το αντίθετο θα δυσχεραίνεται η ζωή των προσφύγων και των μεταναστών. Είναι λάθος το σημείο εκκίνησης όπως σας είπα, στο Συμβούλιο μας λένε ε, ότι θα ε, πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τη σύμβαση της Γενέβης που έχουμε προσυπογράψει και που μας υποχρεώνει να παράσχουμε προστασία σε όσους τη χρειάζονται. Αυτό πρέπει να είναι το σημείο κίνησης και αν ε, χρησιμοποιήσουμε αυτό το σημείο κίνησης οφείλουμε να καταγγείλουμε αυτά που κάνει το Συμβούλιο. Τα κομβικά σημεία, hot spots, την πολιτική επιστροφή, η έννοια της ασφαλούς χώρας, η αύξηση στον αριθμό των κρατήσεων είναι σε αυτές οι πολιτικές. Κανείς δεν τις πιστεύει για τη μετανάστευση, για τους μετανάστευση και τους πρόσφυγες δημιουργεί ακόμη περισσότερα προβλήματα και σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει μελλοντική λύση αυτό. Από την QNGL θέλουμε ε, να ε, δοθεί με περισσότερη έμφαση στην έρευνα και στη διάσωση, μικρότερους ρόλους για τη Frontex και ε, πιο αξιοπρεπής μεταχείριση των προσφύγων. Το Δουβλίνο, κατά τη γνώμη μας, είναι μέρος του προβλήματος. Υπάρχουν και πολλές άλλες προτάσεις που συζητούνται. Ε, και κάποιε είναι καλέ. Ακούσαμε και από τα μέλη του πάνελ για την ε, μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση. Καλέ οι προτάσει του Συμβουλίου δεν ακούν όμω γιατί με αυτά τα στοιχεία η Σουηδία τελικά θα υποδέχεται λιγότερου πρόσφυγε από ό,τι τώρα. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Πρέπει να υπομειστούμε την ευθύνη που, μας, ε, που επιτάσσει η κατάσταση. Χρειαζόμαστε επίσης μετατόπιση σε σχέση με τα σημεία εισόδου. Ε, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση με τη Σύμβαση της Γενέβης, να ε, οφείλουμε να παράσουμε την προστασία που οι άνθρωποι χρειάζονται και αυτό ε, συνεπάγει θα ακολουθήσουμε διαφορετική κατεύθυνση. Κλοντ σε ζητώ συγγνώμη που σας πιέζω, παρακαλώ να υπερβαίνετε τα δύο λεπτά. Ιγνάτσιο e Καρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τις παρεμβάσεις όλων των ομιλητών, ε, συζητήθηκαν διάφορα θέματα και είναι δύσκολο να τα συζητήσουμε όλα σε δύο λεπτά. Επομένως θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ ε, στην... Ε, ε, κίνηση. Ε, γίνεται και μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, πρέπει να το υπενθυμίσουμε, ε, το υπενθύμισαν και οι συνάδελφοι. Σήμερα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, από την οποία θα προκύψει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα θα είναι ερνητική και δεν θα επιλύσει το δράμα αυτών των ανθρώπων. Ε, είναι, δεν χρειάζεται να πω περισσότερο, διότι στο θέμα της μετανάστευσης βγαίνει στην επιφάνεια ο εγωισμός των κρατών μελών, ε, οι εθνικοί ε, εγωισμοί και τα εθνικά συμφέροντα και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ενωμένη ενώπιον ενός θέματος αλλά και μιας εποχής που είναι κατά πάσα πιθανότητα ιστορικής. Ε, πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν ότι η καταπολέμηση των διακινητών είναι μία από τις απόλυτες προτεραιότητες την οποία πρέπει να προωθήσουμε. Ε, αυτά, δεν συνειδητοποιούν το γεγονό ότι οι διακινητέ είναι πολύ πιο πονηροί και πολύ πιο γρήγορα αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Όταν ξεκινάει λοιπόν μια μάχη και προσπαθούμε να διαλύσουμε σκάφη ή να τα βυθίσουμε, ε, οι ίδιοι ε, οι ιδιοκτήτες ε, των σκαφών είναι ε, αυτοί οι οποίοι ε, βάζουν στη θέση τους μετανάστες, βάζουν ένα 15χρονο παιδάκι για παράδειγμα να είναι κυβερνήτης του σκάφους και χάνει αυτό στη ζωή του και όχι ο διακινητής. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να ανατρέψουν την κατάσταση. Θεωρώ ότι η μόνη δράση που πραγματικά θα μπορούσε να βοηθήσει τα πράγματα, χωρίς να παραβλέψω βεβαίως και το γεγονό ότι πρέπει να τροποποιηθούν όλες οι πολιτικές μακροπρόθεσμα, είναι να επιτρέπουμε την νόμιμη πρόσβαση. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε το θέμα των θεωρήσεων, αυτέ τι ανθρωπιστικέ θεωρήσει και να δημιουργήσουμε κατάλληλε προποθέσει για αυτού τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από καταστάσει πολέμου και ε, απειλής, να ζήσουν και να φτάσουν με ασφαλή και νόμιμο τρόπο στι χώρε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι γιατί έχουμε ψηφοφορίες στι 11. Η κυρία Ιώτοβα έχει το λόγο στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μάρτιν και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Κύριε καθηγητά, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς πώς το βλέπετε, 40.000 συν 2.000 ε, που προτείνεται να επανακατασταθούν στα κράτη-μέλη θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κάθε κράτος μέλος, γιατί αναφερθήκατε εκτενώς αυτό. Θα πρέπει επίσης να είναι ε, ένα από τα κριτήρια επανεγκατάστασης οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ο κ. Κέρκοπ, που είναι συντονιστής των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. δεν θα είμαι πάρα πολύ ειδικό. Ακούσαμε, δεν θα πω σε δηλαδή, ακούσαμε μια εκτενή περιγραφή από τους ομιλητές μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και τα επόμενα χρόνια και 10 και 20 χρόνια. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση είναι αποσπασματική και βραχυπρόθεσμη και εδώ εντάσσω και κάποιες πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι προτείνει να κάνουμε με την μετανάστευση το βλέπει αριθμητικά το ζήτημα. Μετράει ανθρώπους και τους διανέμει, που για μένα είναι απολύτως απαράδεκτο μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να το δούμε αλλιώς. Πολύ ευρύτερα και πολύ σφαιρικότερα όλο αυτό το θέμα. Όπως γνωρίζετε, Πρόεδρε, διατέλεσα υπουργό μετανάστευση στη δεκαετία του 90 στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση από τη σημερινή πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν και ορισμένοι δεν θέλουν καν να έρθουν στην Ευρώπη από άλλα μέρη του κόσμου. Ορισμένοι έρχονται με ελεύθερη βούληση δική τους και κάποιοι άλλοι ε, επειδή θεωρούνται ε, εργαλεία αντικείμενα φορείς κλιματικής δραστηριότητας. Ορισμένοι επιθυμούν να συμμετέχουν ε, στην οικονομική επιτυχία της Ευρώπης, ενώ κάποιοι άλλοι έρχονται επειδή έχουν υποστεί ικτρή μεταχείριση και φρικαλαιότητες και ε, εμπίπτουν στην σύμβαση της Γενέβης του 51 και το πρωτόκολλο 67 και έχουν ε, τη δυνατότητα να θεωρηθούν ε, πρόσφυγες ή ετούντες άσυλο. Εμείς δεν κάνουμε διακρίση, η διάκριση που κάνουμε είναι οι αριθμοί. Προσπαθούμε να τους διαιρέσουμε και να τους μοιράσουμε στα κράτη-μέλη είτε αυτό συμφωνεί με τον πολιτισμό, την κουλτούρα τους, τα προσόντα τους, τις συνθήκες τις οποίες έφτασαν, τους οικογενειακούς δεσμούς κτλ. κτλ. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό και δεν πιστεύω ότι είναι ούτε υπεύθυνη ούτε λογική προσέγγιση. Αυτό μπορεί να ικανοποιεί τις ε, συνειδήσεις ορισμένων ή να είναι πολιτική ε, για τα μάτια, αλλά για μένα η μετανάστευση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και θα συζητηθεί και αλλού σήμερα στις Βρυξέλλες. Μάλλον υποπτεύομαι ότι πάλι βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα θα βγει. Για πάλι δεν ασχολούμαστε με τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι ρίζες, οι πηγές, είτε είναι εγκληματικότητα, είτε είναι ε, από σταθεροποίηση, θα πρέπει να λύσουμε το κακό στη ρίζα του. Επίσης, να καταλάβουμε ότι η διάκριση ε, θα πρέπει να γίνει αλλού, όχι εκεί που την κάνουμε αριθμητικά, αλλά να δούμε γιατί έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, ποιοι είναι και τι θέλουν. Ε, η κυρία Αναγκόμες, παρακαλώ μην ξεπερνάτε το δίλεπτο. Ε, ζητώ συγγνώμη, όταν σας άκουσα κύριε Γιόντσεφ, νόμιζα ότι είχα πιστέψει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο migration is not a crime. Δεν είναι έγκλημα η μετανάστευση. Ο πρώτος βασιλεύς της Πορτογαλίας πριν από χίλια χρόνια ήταν από τη Βουργουνδία, πρόσφυγας ο άνθρωπος. Και με κάποια κριτήρια ε, η βασίλισσα Ελισάβετ είναι μετανάστρια. Ε, γιατί η οικογένειά της είναι γερμανικής καταγωγής, αριστοκρατία. Δηλαδή η μετανάστευση δεν είναι έγκλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Και χρειάζονται νόμιμοι διαβληλεοφόροι για τη μετανάστευση. Μπορεί να μην είναι αυτό το βραχυπρόθεσμο που λέτε που κάνουν κυβερνήσει. Μακροπρόθεσμη χρειάζεται στρατηγική θεώρηση και ευφυής, όπω είπε ο Καθηγητή Μάρτιν. Και βεβαίω χρειαζόμαστε τρόπου να φτάνει ο κόσμο νόμιμα. Αυτό ακριβώ δεν κάνουν τα κράτη-μέλη. Ε, έχουν βγάλει εκεί μια μικρή γαλάζια κάρτα που δεν φτάνει σε καμία περίπτωση και είναι τελείως ακατάλληλη ως μέτρο. Βέβαια τίθεται και το θέμα των προσφύγων και των ετούντων άσυλου. Και ευχαριστώ για αυτά που λέτε. Και θα πρότεινα υπηρεσίες πληροφοριών και οι αστυνομία ή συνοριοφύλακες να πηγαίνουν τρεις μέρες σε ένα καταβλισμό προσφύγων στην Τουρκία για σεμινάρια που έχω πάει εγώ. Όχι αυτά τα πολυτελή, υπάρχουν και στρατόπεδα σκληρά ε, με σκηνές κάτω από τον ήλιο. Ή στο Βόρειο Ιράκ πηγαίνετε εκεί για επιμόρφωση τρεις μέρες και θα καταλάβετε ότι ο κόσμος θα κάνει ό,τι μπορεί τα δύνατα δυνατά για να φύγει από εκεί και να έρθει κάπου αλλού στην Ευρώπη θα βοηθήσει αυτό να καταλάβετε τις προκλήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Μπάουερ που αναφέρθηκε στην Αίγυπτο, γιατί εδώ όλοι συζητάμε για τη Λιβύη, όπου η κατάσταση φυσικά είναι χαόδης και ήταν σκέτη καταστροφή η κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων. Έτσι κι αλλιώς και επικαντάφη ήταν στους καταβλισμούς, αλλά ποιο έδινε τότε δεκάρα. Ε, μου άρεσε αυτό που είπατε για την Αίγυπτο και το ρόλο Τη ίδια της Αιγύπτου στην οργάνωση και τη διακίνηση. Έχω όμω την εξή ερώτηση και ευχαριστώ κύριε Μάρτιν και κύριε Βυζαντίνη για ε, αυτά που είπατε για τα οικονομικά. Και η Ευρώπη κατά τα άλλα παράγει μετανάστες με την πολιτική λιτότητα. Μάρτις είναι η χώρα μου και μάλιστα καταρτισμένους και ειδικευμένους. Και ρωτώ τον καθηγητή πήρες. ναι, Άννα, έχεις Φτάνει στα τρία λεπτά τώρα. Ναι, αλλά πρέπει να το ρωτήσω, γιατί το ρώτησα και χθε την κυρία Μογκερίνη. Για ποιο λόγο η unaf δεν έχει ως πρώτο στόχο το να σώζει ζωές, διότι αυτό είναι υποχρέωση. Όχι μόνο βάσει του δικαίου της θάλασσας, αλλά και από Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Θα μπορούσατε λίγο να επεκταθείτε για τον κανονισμό που χρειάζεται να μην είναι μόνο μια στρατιωτικοποιημένη επιχείρηση, που θα τη βρούμε μπροστά μας ή θα γίνει μπούμεραγκ. Θα πρέπει η θα γινει boomerang. θα πρεπει η ευρωπη να αφιερώνει όλους τους πόρους και τους στρατιωτικούς ε, στη διάσωση ζωών και στο τερματισμό της διακίνησης. Κοίτα, Άννα και συνάδελφοι, αγωνιώ στις 11 ψηφίζουμε και θέλω να προλάβουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας, μην κάνετε. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε για την αυτή μεγαλειότητα. Η κυρία Μουσολίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα πολύ ε, καλές παρεμβάσεις αλλά και προκλητικές ε, συνάμα. Προσκαλέσατε εδώ τον πρέσβη της Ελβετίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος αναφέρθηκε σε 2.000 μετανάστες, δεν ξέρω σε πόσο χρονικό διάστημα. Εμείς υποδεχόμαστε 2.000 μετανάστες τη μέρα. Από αυτά που άκουσα λοιπόν, δεν υπάρχει πλέον η Ευρώπη με τα σύνορα, με τίποτα. Υπάρχει μια άλλη Ευρώπη. Συζητούμε μια άλλη Ευρώπη ε, πλήρως ανοιχτή, με νόμιμες διάβλους και νόμιμη μετανάστευση η οποία όμως δεν είναι η σημερινή Ευρώπη, γιατί υπάρχει μια καλή Ευρώπη και μετά υπάρχει Ευρώπη η οποία χτίζει συνικά τείχη, διότι τα κατασκευάζει αυτά τα τείχη. Επομένως υπάρχουν χώρες α κατηγορίας και χώρια β ε, κατηγορίας. Και έπρεπε να πω στον κύριο Μπάουερ για αυτό το δραματικό ταξίδι που έκανε. Δεν έπρεπε να τελειώσετε το ταξίδι σας εκεί. Το δεύτερο σκέλος έπρεπε να έρθετε να το κάνετε στην Ιταλία. Γιατί στην Ιταλία θα βλέπετε τη χώρα που υποδέχεται αυτούς τους μετανάστες. Υπάρχει ένας αρρωστημένος ιστός Έχουμε τους διακινητές ανθρώπων και μετά στην Ιταλία έχουμε τους εμπόρους ανθρώπων. Κάθε δομή, ε, το έχω πει και σε πιο περιορισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής, Κάθε δομή ε, για 30 μετανάστες παίρνει 85.000 ευρώ ε, το μήνα. Αυτό είναι 900.000 ευρώ το χρόνο. Πρόκειται λοιπόν για μια τεράστια διακίνηση στην πραγματικότητα. Ε, αυτό συμβαίνει στην Ιταλία. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι οτιδήποτε γίνει στη συνέχεια γίνεται τμήμα ενός εγκληματικού συστήματος που αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα οργανωμένο. Δεν υπάρχει μόνο η μαφία, η της Αιγύπτου, έχουμε και την εσωτερική μας. Πρόκειται λοιπόν για θέματα τα οποία συζητώνται εδώ και δεν έχουμε καμία συνέχεια στη συνέχεια. Πολύ ωραία νόμιμη μετανάστευση, δεν χρησιμεύει σε τίποτα να ε, καταστρέψουμε του ε, Να πάμε, να πάρουμε του μετανάστε με κρουαζιερόπλαιο. Δεν είναι πρόκληση να έρθουν με τα κρουαζιερόπλαια και μετά να, ε, να, για να του σώσουμε να μην πέφτουν θύματα των σκαφών. Και μετά τι θα του κάνουμε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, άκουσα μια σειρά από ομιλίε που πραγματικά με εκπλήσουν, διότι αν έστω από εμά είχε είχε κάνει αντίστοιχη ομιλία στην Ιταλία θα είχε κάτι αντιδράσεις πάρα πολύ αρνητικές. Πραγματικά λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε για αυτούς τους αρεστημένους ιστούς που υπάρχουν στις χώρες υποδοχής. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και προκαλούν και συγκινήσεις, αλλά δυστυχώς μας περιορίζει ο χρόνος μας και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Εμίλ Ράντευ στη συνέχεια. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. «170 εκατομμύρια ευρώ έκανε οι διακινητές κέρδος το 2014. Πρέπει να κάνει κάτι αμέσως η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, η UNAFOR, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εάν περιοριστεί μόνο στην καταστροφή και διάλυση σκαφών σε διεθνή ύδατα και στη Λιβύη. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από τους διακινητές ε, στη Λιβύη και από άλλες ε, χώρες ε, συνεργάζονται με εμπόρους ε, που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ε, τους διευκολύνουν να περνούν αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τις διάφορες χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, για τις ε, δυνάμεις επιβολής του νόμου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργάζονται ώστε να μπορέσουν να καταπολεμήσουν ε, το φαινόμενο και να πατάξουν αυτά τα εγκληματικά δίκτυα. Έχουμε κάποια παραδείγματα. Στη Βουλγαρία η αστυνομία κατάφερε να αντιμετωπίσει μια οργάνωση από την Τουρκία και ελπίζω να έχουμε και κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσπαθήσω να τα πω σε ένα δίλεπτο. Να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους ομιλητές ε, που ε, αναφέρθηκαν σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ τον Υπουργό Γιόντσεφ. Ε, ήταν πολύ γενναίες οι προτάσεις τους και καθόλου κομφορμιστικές. Ευχαριστώ και τον πρέσβη, τον κύριο Μπαλτσαρέτη, για την παρουσίασή του, που είπε ε, ποιες είναι οι εθνικές ευθύνες. Ότι δεν είναι κούφια λόγια, είναι γεγονός, οι ευθύνε είναι στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση. Άλλο η μετανάστευση ε, άλλο η λάθρο μετανάστευση, άλλο οι πρόσφυγες, άλλο οι οικονομικοί μετανάστες. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και θα πρέπει επίσης να σεβόμαστε και την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών μας. Η οικονομική μετανάστευση είναι κάτι ε, το οποίο δεν μπορούν να αντέξουν πολλές οικονομίες στα κράτη-μέλη μας. Υπάρχουν χώρες όπως η Βουλγαρία ή η Λιθουανία Φερρυπίν όπου πάνω από 10% του πληθυσμού έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Και υπάρχουν μεγάλες ε, περιοχές ε, με υψηλή ανεργία ή μεγάλες περιοχές ε, που έχουν εγκαταλειφθεί από τον πληθυσμό. Αυτό οφείλεται στην πτώση του οικονομικού σιδηρού παραπετάσματος κάθε χώρα θα πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της με διμερείς συμφωνίες. Βεβαίως και χρειάζεται αλληλεγγύη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά θα κάνει να ασχολείται με τις δικές της αρμοδιότητες. Ε, στην Ευρώπη έχουμε ε, πολλούς εσωτερικούς μετανάστες, πολύ μεγάλες ανισότητες και δικά μας ζητήματα που χρειάζεται να λυθούν. Η ε, κυρία Κριστίν Ρεβονταλόν, τελευταία ομιλήτρια σε αυτό τον κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για τις παρεμβάσεις σας που καταδεικνύουν ότι έχουμε δύο οικονομικές λογικές οι οποίες συγκρούονται στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η μετανάστευση στην Ευρώπη. Αυτοί που σήμερα προκρίνουν τα κράτη-μέλη λέγει ότι δίνουμε πολλά κονδύλια για την καταστολή των δικτύων των διακινητών προφανώς και την αστυνομική διαχείριση των μεταναστών, ε, την ε, επαναπρόθεση τους στα σύνορα αυτά έχουν ένα οικονομικό κόστος και θεωρείται η μετανάστευση ως πρόβλημα, ως πίεση. Αυτά ακούμε και ως έννοιες και ως όρους. Και υπάρχει και ο άλλος τρόπος και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μάρτιν και τον κύριο Βετζεντίνη για τις παρουσιάσεις όπου αποδεικνύουμε ότι η μετανάστευση έχει μια πραγματική οικονομική υπεραξία. Το γνωρίζουμε αυτό. Στη Γαλλία βλέπουμε ότι η μετανάστευση αποδίδει και είναι πολύ περισσότερα αυτά που αποδίδει από όσα κοστίζει. Όλοι θέλουμε να έχουμε μια συνολική θεώρηση και αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Να δούμε και την οικονομική και την νόμιμη μετανάστευση. Είναι πολύ εύστοχο αυτό. Θα πρέπει να σταματήσει η σαλαμοποίηση για τις γαλάζιες κάρτες ε, ε ανειδίκευτοι ή ειδικευμένοι. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι κύριε Βιντσεντσίν. Τι γίνεται με τους κλάδους της απασχόλησης που ε, ψάχνουν ένα εργατικό δυναμικό και ανειδίκευτο καμιά φορά ε, και δεν βρίσκουν. Κύριε Μάρτιν, είπατε ότι στο μέλλον θα χρειαστούμε εκατομμύρια μετανάστες. Ξέρουμε ήδη από τώρα ε, ποια θα είναι η δημογραφική εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Φυσικά και θα χρειαστούμε μετανάστες και να ξεφύγουμε από αυτή την ε, χήμερα την ψευδέστηση ότι είναι κόστος. Είναι και οικονομικό ζήτημα και τα οικονομικά ζητήματα εξετάζονται κατά προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ Κριστίν. Λοιπόν, τώρα στους ομιλητές έρχομαι. Δεν θα σας δώσω χρόνο. Θα πρέπει εσείς να αποκρισταλώσετε τι ερωτήσεις έγινε σε εσάς για να απαντήσετε. Κυρίως τις ερωτήσεις των βουλευτών και λιγότερο τα σχόλια για να απαντήσετε. Και αν υπάρχουν ιδιαίτερες ερωτήσεις ή δεν ικανοποιηθούν οι συνάδελφοι από την απάντηση, μπορούμε να έχουμε και γραπτή απάντηση. για το καλέ ας πούμε ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται εκεί και με τα νομικά ζητήματα αλλά θα ρωτήσω τον καθηγητή Πίερς αργότερα. Λοιπόν, ο ε, κύριος Γιόντσεφ δύο λεπτά το πολύ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να υπάρχουν και νόμιμοι διάβλοι μεταναστευτικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι απολύτως πεπισμένο ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικέ ροέ. με μια συστηματική ολιστική προσέγγιση. Έτσι μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα μεταξύ των οποίων και αυτά που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Παρακαλώ να μην παρανοήσετε αυτά που λέω. Δεν είναι ότι δεν τους θέλω αυτούς τους ανθρώπους και πιστεύω δεν πρέπει να τους θέλουμε. Τους, ε, εκεί ήμουνα και τους έχω κοιτάξει στα μάτια και νιώθω τα βάσανα που υπομένουν και ξέρω ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους. Όμως μεταξύ αυτών υπάρχουν και πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Έχω πολλά τέτοια παραδείγματα. Εάν δεν μπορέσουμε να, χωρίσουμε, να διαχωρίσουμε, να διακρίνουμε αυτούς τους επικίνδυνους ανθρώπους από αυτούς που χρειάζονται βοήθεια, τότε θα υπάρχει μεγάλη απειλή για τα δικαιώματα όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Αν σας ζητήσω να σηκώσετε ένα τόνο, δεν μπορείτε. Ε, είναι θέμα πόρων. Είναι θέμα διοικητικών δυνατοτήτων. Προσοχή Μήπως ξεφύγει, μας ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο και τότε θα υπάρχει κίνδυνος για όλους μας. Ευχαριστώ. Κλοντ Μορές, ξέρω ότι θέλετε να μας πείτε πολλά περισσότερα, αλλά είναι δύσκολη κατάσταση και ξαναλέω, όσοι θέλετε να ρωτήσετε περισσότερα τον κύριο Στόσγεφ, να τους επικοινωνήσετε δημερός. Κύριος Μπάουερ, πάλι δύο λεπτά. Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Γόντσεφ. Νομίζω είναι ψευδέστηση να ψηφ... νομίζουμε ότι θα μπορούσαμε με την πολιτική που ακολουθούμε μέχρι τώρα να αποτρέψουμε να, να έρχονται και επικίνδυνοι άνθρωποι με τους πρόσφυγες, dangerous people όπως τους είπατε. Ε, ε, εάν νομιμοποιούσαμε τη μετανάστευση με τον τρόπο που προσπάθησα να περιγράψω προηγουμένως, θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε πολύ περισσότερο το ποιος έρχεται και ποιος δεν έρχεται. Τώρα δεν τους ξέρουμε γιατί έρχονται όλοι οι παράνομα, περνάνε κάτω από το ραντάρ και είναι αστυνομική ψευδέστηση να νομίζουμε ότι με περιορισμούς αποτρέπουμε τέτοια φαινόμενα να έρχονται και οι εγκληματίες και ότι δήθεν προστατεύεται οποιοδήποτε. Είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να αποφύγουμε οι άνθρωποι αυτοί να ε, μπαίνουν καν σε αυτά τα σκάφη. Στα λιμάνια της Λιβύης είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρωπιστικούς διάβλους, διαδρόμους για να φέρνουμε στην Ευρώπη τους πρόσφυγες, ε, που είναι πρόσφυγες πολέμων, επαναλαμβάνω, όπως έγινε με τη Βοσνία. Για την Ιταλία, με ρωτήσατε, είναι σκάνδαλο φυσικά αυτό που συμβαίνει και στην Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου, έχει αφήσει στη μοίρα της περίπου την Ιταλία και σύμφωνα με τις δικές μου εμπειρίες, ε, η Ιταλία μποϊκοτάρει το ε, Δουβλίνο. Πήγα και εγώ στην Ιταλία, είδα και πρόσφυγες εκεί, τους οποίους αμέσως άφησαν ελεύθερους οι αστυνομικέ αρχές για να προχωρήσουν στην Ευρώπη χωρίς να γίνει δακτυλοσκόπηση. Ε, τρεις συνάδελφοι που ήταν, φίλοι που ήταν ε, μαζί μου ε, προσπάθησαν να τους βοηθήσω να πάνε στη Στοχόλμη, στη Σουηδία και με πιάσανε στην Αυστρία, με συνέλαβαν ως διακινητή. Ε, Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος που βοηθάει κάποιον ανθρωπιστικά ε, να φύγει ως πρόσφυγας από κάπου που κινδυνεύει η ζωή του, αν μπορεί να χαρακτηριστεί διακινητής. Εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι τώρα στη φυλακή γιατί προσπάθησαν να βοηθήσουν μέλη της οικογένειας να περάσουν τις Άλπεις από την Ιταλία προς τη Γερμανία και ε, χαρακτηρίστηκαν διακινητές και φυλακίστηκαν. Θυμίζω το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας DDR. Και εμεί στη Γερμανία έχουμε, είχαμε τείχο. Τώρα όπως ε, αρχίζει να ε, γίνεται στην Ευρώπη γύρω-γύρω, εκατοντάδε ήταν οι νεκροί στις τέσσερις δεκαετίες ε, ζωής αυτού του τείχου. και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι είμαστε ανώτεροι ηθικά από το καθεστώς της DDR, αλλά ταυτόχρονα αφήνουμε 20.000 ανθρώπους να πνίγονται στα εξωτερικά μας σύνορα. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω. Δεν πρόκειται να μπω σε ζητήματα ασύλου και ανθρωπιστικών διάβλων, γιατί τα, τα ακούσαμε όλα από τους συναδέλφους. Δύο ε, θέλω να κάνω για την μπλε κάρτα και για τους τομείς όπου χρειαζόμαστε νόμους μετανάστες. Για την οδηγία, για την μπλε κάρτα. Φοβερή ε, ψευδιέστηση και αποτυχία διότι ο στόχος της οδηγίας ήταν να επιλεγούν μετανάστες επί τη βάση των δεξιοτήτων τους και να προσελκύσουν ε, ε, εξειδικευμένους και μόνο μετανάστες. Μα απέτυχε διότι δεν χρειαζόμαστε μόνο αυτούς και λίγους τέτοιους χρειαζόμαστε σε σχέση με τους περισσότερους που χρειαζόμαστε ε, με άλλα επίπεδα ειδίκευσης και σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας. Αν πραγματικά θέλουμε να θεωρήσουμε την οδηγία για την μπλε κάρτα τότε δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με το μισθό αυτών των ε, εργαζομένων. Όταν αναφερόμαστε στα 1500 ευρώ μισθό, και το μέσο μισθό που θα πρέπει να παίρνουν αυτοί οι μετανάστες δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό μισθό. Δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτό το κριτήριο για να γίνει επιλογή των μεταναστών σε σχέση με άλλους που επίσης είναι μέλη της αγοράς εργασίας. Δεν είναι το πρόβλημα ο μισθός. Το πρόβλημα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο ε, ε ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση, χρειαζόμαστε και άλλα επίπεδα ειδίκευσης σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας. Έχουμε πολλές κενές θέσεις σε άλλα επίπεδα και σε άλλους τομείς. Και έχουμε να λύσουμε το θέμα της ανεργίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από αυτό των μεταναστών. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε τις οικονομικές επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας χωρίς τους μετανάστες. Χωρίς αυτούς δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα το σύστημα ιατρικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης λόγω της γύρανσης του πληθυσμού. Πέρα από τη δημογραφική πτύχη, χρειαζόμαστε διαφορετική βασικά στοιχεία που πρέπει να συνυπολογιστούν για να καταρτήσουμε μια προσέγγιση. Θα πρέπει να θεωρείται προσθέμενη αξία και θετική συμβολή η μετανάστευση. Όχι μόνο για την αγορά εργασίας, γενικότερα όμως για την κοινωνία. Ευχαριστούμε ο καθηγητής Μάρτιν. Ευχαριστώ. Πέντε πράγματα σε δύο λεπτά. Καταρχάς, για την μπλε κάρτα ποτέ δεν θεωρήθηκε ως μέσο μετανάστευσης ε, για λόγους εργασίας. Ήταν ένας τρόπος να προσελκύσουμε διεθνή ταλέντα. Και αυτό ήταν για να βοηθήσουμε τις πολυεθνικές εταιρείες. Χρειάζεται. Καλό είναι να το κάνουμε, αλλά να το έχουμε, αλλά ε, δεν έχει σχέση. Ε, μπορώ να σας πω και περισσότερα από αυτού. Δεύτερο θέμα, το θέμα της αντικατάστασης. Να είμαστε βέβαιοι ότι μετανάστες από ε, τρίτες χώρες δεν θα αντικαταστήσουν το εργατικό δυναμικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει σχέση μεταξύ ενδοκινοτικής κινητικότητα και διεθνή πολιτική μετανάστευση. και επίση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νόμιμοι μετανάστες θα ε, εργάζονται ε, με τις ίδιες συνθήκες και θα λαμβάνουν τους ίδιους μισθούς ε, με τους Ευρωπαίους. Αυτό ισχύει σε κάποιες χώρες, όχι τόσο αποτελεσματικά σε άλλες και να υπάρχει ε, ένα ευρωπαϊκό τεστ για την αγορά εργασίας που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα νέο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, το δημογραφικό θέμα. Ε, το ανέφερα και στην παρουσίασή μου, έχουμε τα στοιχεία, είναι σαφέστατα τα στοιχεία και μάλιστα σε μία ε, έκθεση που ετοιμάζει το Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής ετοιμάζεται μια έκθεση που περιλαμβάνει μια αναθεώρηση όλων των μελετών που έχει γίνει και σε αυτή την περίπτωση δεν θέλουμε μόνο υψηλών δεξιοτήτων ε, ε, μετανάστες αλλά χρειαζόμαστε και ε, προσωπικό χαμηλότερων προσόντων και επίσης χρειαζόμαστε και γυναίκες στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά την ερώτησή σας ε, για τις ποσοστώσεις επανεγκατάστασης για τους ετούντες άσυλο, όσα κριτήρια θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μπορείτε να αξιολογήσετε τεχνικά το κάθε κριτήριο. Αλλά υπάρχει το εξή πολύ σαφές θέμα. Ε, στη χώρα μου, νομίζω ότι μπορώ να το πω εγώ, ε, η, Ισπανία είναι μία από τις χώρες που λέει ότι θα πρέπει να περισσέξετε περισσότερο την αγορά εργασίας γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία. Ναι, μεν, αλλά είναι και λίγο υποκριτικό σε μια χώρα με 5,5 εκατομμύρια ανέργους να λέμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε 5.000 ετούντες άσυλο γιατί είναι έτσι η κατάσταση στην αγορά εργασίας ε, και οι περισσότεροι από αυτούς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ναι μεν, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό επιχείρημα αυτό το επιχείρημα. Επίσης, ένα ουσιαστικό ζήτημα που μπορώ να σχολιάσω ακόμα πρέπει να ε, ξεπεράσουμε αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών μετανιστών. Είναι υποκριτικό να χρησιμοποιούμε αυτή τη διάκριση γιατί υπάρχει ένα σύστημα διεθνούς προστασίας. Από ηθική σκοπιά, άνθρωποι οι οποίοι πεινούν και έχουν ανάγκες ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν προστασίας. Και αν τα κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο, ε, πέραν των νομικών υποχρεώσεων για την ε, διεθνή προστασία, θα ήθελα να λάβετε υπόψη και τη διεντολογική σκοπιά, την ηθική υποχρέωση. Ο καθηγητής Πίερς. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα μου έθεσαν άμεσα και θα ασχοληθώ με αυτά. Η κυρία Βίξτρον πρώτα απ' όλα με ρώτησε για τις δημογραφικές τάσεις και τη μετανάστευση. Φυσικά ε, πρόκειται πρωτίστως για εθνική αρμοδιότητα και μόνο συμβουλές μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επιδόματα, για τα παιδιά, για επιδόματα που δίνονται μέσα από την εργασία, ούτως ώστε η αγορά εργασίας να υπάρξει η αντιστήξη ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις οικογενειακές ανάγκες. Άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας, ε, το Συμβούλιο θα διαπραγματεύεται με το Κοινοβούλιο, θα δούμε τώρα αν θα υπάρξει συμβασμό. Υπάρχουν ε, δύο τομεί όπου η Ένωση θα μπορούσε να επέμβει αμεσότερα. Η οδηγία για την μπλε κάρτα είχε γίνει μια πρόταση για νεότερους ανθρώπους. Ε, ίσως θα έπρεπε να επανέλθει αυτή η πρόταση με την αναθεώρηση της οδηγίας για την μπλε κάρτα και όπως είπε και ένας άλλος ομιλητής, αυτή η οδηγία δεν πρέπει απαραίτητα να καλύπτει μόνο την υψηλή ειδίκευση. μπορεί να καλύπτει γενικότερα τα κενά ως προς τις ειδικότητε. Δηλαδή όπου υπάρχει ένα κοινό μπορούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία φυσικά με ευνοϊκούς κανόνες για την οικογενειακή επανένωση. Δεύτερο τομέας όπου μπορεί για τη μετανάστευση να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δική σας πρόταση για τους φοιτητές και τους ερευνητές με αυτή τη χρήσιμη ρήτρα στο τελικό κείμενο για την ενθάρρυνση των φοιτητών να παραμείνουν μετά την απόκτηση πτυχίου. Δηλαδή καλό θα ήταν, πολύ χρήσιμο, αυτοί που φίτησαν εδώ να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι αρκετά νέοι ούτως ώστε να εργαστούν ολόκληρη τη ζωή εδώ και να ε, δημιουργήσουν οικογένεια. Ε, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με τις απαιτήσεις για την μακρά διαμονή. Η Γιουνάφο, κυρία Γκόμε, ε, δεν νομίζω ότι είναι δυνατό με την κατάσταση στη Λιβύη, ούτε και νόμιμο, διότι ε, η νομική υπηρεσία θα, ε, το, θα ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή πρόκειται για εξωτερική πολιτική. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να σταματήσετε το Συμβούλιο. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ε, επιδιώξετε μεγαλύτερη λογοδοσία ε, για αυτά που κάνει το Συμβούλιο. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριος Κλόντ Μονές, ε, για την πίεση που σας ασκώ τώρα. Βλέπω και κοιτάζω τις συνεισηγήτριες, γιατί έχουμε και τη Δευτέρα Ιουλίου ως προθεσμία η Ρομπέρτα και η Σισίλ. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Είναι πάρα πολλές οι θέσεις που ακούστηκαν εδώ στην Επιτροπή μας. Για να συμπεράνω, συμφωνούμε όλοι ότι η προτεραιότητά μας είναι να σώζουμε ζωές και να προστατεύουμε τους ανθρώπους αυτούς που αξίζουν και χρειάζονται προστασία. Όμως ε, χρειάζεται και ε, ισορροπία. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος κάθε χώρας και οι δυνατότητες απορρόφησης που έχει. Και ε, οι άνθρωποι που χρειάζονται προστασία ε, θα πρέπει να την έχουν με κάποια διαφοροποίηση. Και εδώ ρωτάω τον κύριο Πίερς να δούμε, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της ανθρωπιστικής θεώρησης διαβατήριου. Λοιπόν, προτεραιότητα να μην αφήνουμε κανένα να πέσει στα νύχια των διακινητών και να προστατεύουμε τις ανθρώπινες ζωές. Και όσοι πιστεύουν ότι ε, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα αν δεν αντιμετωπίσουμε τους διακινητές, έχουν και εκείνοι το δίκιο τους, αλλά οι διακινητές δεν είναι ε, διασώστες, δεν είναι σωτήρες, δεν τους νοιάζουν οι ζωές των ανθρώπων αυτών. Το κέρδος τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει να πνίγονται, να δεν πνίγονται οι άνθρωποι. Αυτό θα πρέπει να τερματιστεί. Ευχαριστώ, Ροπέρτα. Η Σεσίλ, ένα τελευταίο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους και συζητητέ για τη συνεισφορά τους ε, και για τα όσα μας είπαν ε, και τους ομιλητές. Ε, συμφωνώ ε, με αρκετές από τις έννοιες και πολλά από αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι πολύ σημαντικό από πολιτικής αλλά και πολιτισμικής σκοπιάς κατά την άποψή μου, το οποίο αναφέρθηκε στην ε, ε, παρουσίαση του κυρίου Μάρτιν και του κυρίου Βισεντίνη. Πρέπει να γίνει μια ριζοσπαστική αλλαγή και σε θέματα ορολογίας, διότι αναφερόμαστε σε μετανάστες χωρίς έγγραφα που δεν είναι ούτε παράνομοι ούτε κλιματίες. Επομένως, όταν αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε περί ποιου πράγματος ομιλούμε, σίγουρα θα μπορέσουμε να νομοθετήσουμε καλύτερα και να ρυθμίσουμε όλο τον τομέα. Ευχαριστώ τον κύριο Μπάουερ για την εμπειρία του, διότι χρειαζόμαστε και μια ανθρώπινη εικόνα σε αυτά για τα οποία νομοθετούμε. Και η του είναι πάρα πολύ χρήσιμο, για κάποιον ο οποίος ε, βλέπει λίγο πιο ε, απομακρυσμένα, από πιο μακριά αυτά τα επεισόδια και δεν έχει μια πραγματική εικόνα της κατάστασης. Κάτι τελευταίο, το, στο οποίο θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε, ε, Κύριε Πύρης, θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι για τις θεωρήσεις έχω την εξή ερώτηση. Ποιο θα πρέπει να είναι το νομικό πλαίσιο ε, βάσει των οποίων θα μπορούσαμε να έχουμε μια νέα πολιτική για τι ανθρωπιστικέ αυτέ θεωρήσει ε, στην νομοθεσία για τι θεωρήσει. σω τι επόμενε μέρε θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ, Σεσίλ. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ και του συναδέλφου ουσιαστικότατη συζήτηση σήμερα το πρωί για τη συνολική και σφαιρική θεώρηση. Η επόμενη συζήτηση για την έκθεση αυτή είναι στις 2 Ιουλίου. Σα ευχαριστώ πολύ για τους ομιλητές και τους συναδέλφους. So colleagues, we proceed to the votes. Um... Προς uh, τις ψηφοφορίες οδεύουμε. Αμέσως μόλις καθαρίσει εδώ το πάνελ.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 Colleagues, take your seats. Um, we're going to proceed to the vote. Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι, ακολουθούν ψηφοφορίες. Okay, we proceed to the first vote. Λοιπόν, προχωρούμε. Πρώτη ψηφοφορία. Εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν Προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση για την Αναγκαστική Εργασία τη ΔΟΕ σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει. Η σύγκεντρια είναι η κυρία Χέλγα Στέβενς. Μία και μοναδική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Υπάρχει κανείς που να μην έχει την κάρτα του. Μπράβο, Ζεράρ. Άλλος, είστε όλοι έτοιμοι. Η Άννα, όχι. Διαδικαστικό έχετε. Όχι, δεν είναι διαδικαστικό. Κυρία Σίπελ, δεν έχω ακόμα την κάρτα μου, την ηλεκτρονική, απλώς κοιτάξτε το χέρι μου. Αυτό δεν είναι διαδικαστικό. Αυτό είναι σφάλμα στην οργάνωσή σου. Ωραία. Λοιπόν, ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες μετράμε ένα χέρι και είναι και συντονίστρια. Πω, τη σκέτη απογοήτευση. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Okay, colleagues, the Audi... Okay. Λοιπόν, περισσεύει ένας φιλελεύθερος. Μπορείτε παρακαλώ να αφαιρέσετε τον υπεράριθμο. Ένα τακτικό μέλος κιόλας. Εντάξει. Εντάξει. Η Άλντε έχει αφαιρέσει τον υπεράριθμο. Εδώ δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Εντάξει, εντάξει, μην ενισχύετε. Πέρας ψηφοφορίας και θα σας πούμε. Ένα χέρι μετράμε στους σοσιαλιστές και ένα μηχάνημα που δεν λειτουργεί. Συν δύο δηλαδή σοσιαλιστές και δημοκράτες που δεν ψηφίζουν ηλεκτρονικά και τους προσθέτουμε. Διανατάσσεως χειρός. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας κυρία Χέλγα Στέβενς. Προχωρούμε στην επόμενη ψηφοφορία. Συνάδελφοι, 30 και 31η ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Τραϊάν Ουγκού Ρεάνο είναι ο εισηγητής. Και ψηφίζουμε πρώτα την τροπολογία υπαριθμών 3. Όλα ηλεκτρονικά. Όχι. Η 3 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Η τροπολογία περιφών 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται, διορθώνει ο πρόεδρος. Η τροπολογία περιφών 5. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ συνάδελφοι να σηκώνετε χέρια για να σας βλέπω. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 3. Συμβαστική 3. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 7, τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά απόχες, εγκρίνεται, συμβαστική ήταν αυτή. Η τροπολόγια 13 υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Η 14 υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. Η τροπολογία υπέρ 15 υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Η 17 υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ γιατί δεν είναι σαφές είμαστε στη 18 άρχεται ηλεκτρονική επαλήθευση πέρασε εγκρίνεται τροπολογία 19 ψήφι υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 20 υπέρ όχι 21 διορθώνει πρόεδρος 21 ειπέ. κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην τελευταία έκθεση. We move to the, um, Λοιπόν, σχέδιο ψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια. Συμβιβαστική 1. Α, όχι, μισό λεπτό, συνάδελφοι. Ολόκληρη ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Ναι. Ε, εκτός από κάποιους που δεν έχουν τις ηλεκτρονικές κάρτες μαζί τους, θα μας πούνε πώς ψηφίζουν. Άλλος κανείς. Α, ήρθε λέει κυρία Σίπελ, ωραία. Και δουλεύει και το μηχάνημα. Δουλεύει εσύ, όχι εσύ η κάρτα σου. Εντάξει. Όλα τα μηχανήματα δουλεύουν και οι κάρτες είναι εδώ. Ε, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για την πρώτη συμβαστική. Παρακαλώ. Πέρασε. Τροπολογία 41. Παρακαλώ. 41. 41. σαράντα ένα, ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε.

Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 53 σε τμήμα, ε, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 53 το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 56. Ψηφίζουμε για το τελευταίο τμήμα. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 58. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 59 το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 59 το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 62. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε μόνο. Παρακαλώ. Πέρας. Κρίνεται. 69. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 70. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 71. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 72. Αυτή είναι συμβατή με την 49. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 73 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πρέπει να σας το διαβάσω Το πρώτο τμήμα, όλο το κείμενο και βγάζουμε ε, υπό την πρόφαση της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Ε, ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Παρακαλώ. Για το πρώτο τμήμα. Θέλετε να σας το ξαναδιαβάσω. Όχι, για την 73 της Τζούδης Ατζεντίνη. Κατά τμήματα ψηφοφορία από το ΕΛΚ. Το πρώτο τμήμα, ολόκληρο το κείμενο χωρίς τα ακόλουθα. Ε, με την ε, ε, πρόφαση του, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ιδιαίτερο. Ζητώ συγγνώμη. Εγώ έκανα λάθος. Εντάξει, ωραία. Για το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε τώρα. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Για το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 74. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 75. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 81 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 84 ψηφίζουμε. Ξέχασα να σας πω ότι ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα στην 84. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Γκρίνεται. 94. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Διορθώνει ο πρόεδρος. Όχι συμβαστική 7. Πάμε στην 108. Ψηφίζουμε. Πιστεύω να, να κάνουμε το παράδεκτο και να περάσει. Πέρας. Απορρίπτεται. 109. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 111. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 112. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 113. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 114. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 8. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. τροπολογία 117 άρχεται ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 122, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 123 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Με το Strongly the issue of migration, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Το υπόλοιπο κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 124. Α, συγγνώμη συνάδελφε, συμβαστική τροπολογία 10. Α, όχι, σωστά. Είχα δίκιο, είχε κάνει λάθος η γραμματεία, σημειώστε το. Βελτιώνουμε. 124. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10, άρχια της ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 131, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 132. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 138, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 139, άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 κατά τμήματα κατόπιν αιτήματος των πρασίμων πρώτο τμήμα agrees μέχρι stakeholders. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα από το calls for bolder μέχρι το propaganda. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 148. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 149. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της εγκρίνεται. 151. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 157. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 159 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 160 κατά τμήματα πρώτο τμήμα recalls μέχρι groups. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 161. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 162. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εκρίνεται. 164. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 165. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 167. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 170. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Τώρα. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 175. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 173, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 176, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας πληροφορίας. Εγκρίνεται. 177. Άρχεται πληροφορία. ψηφοφορία. Πέρας πληροφορίας. Εγκρίνεται. 178. Άρχεται πληροφορία. ψηφοφορία. Πέρας πληροφορίας. Εγκρίνεται. 179. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 150. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα Στι αιτιολογικέ εξηγήσει. Τροπολογία 1, άρχεται ψηφοφορία. αναφορέ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 κατά τμήματα κατόπιν ετήσεως του ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Άνα πρέπει να ψηφίσεις. Τροπολογία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε σε τηλεολογικές σκέψεις. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 19, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 33 απορρίπτεται. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Αρχίσαν και εμένα και με ενοχλούν τα διάχτυλά μου από το πάτα-πάτα. Εγκρίνεται και αυτό. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Has everyone Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μικρή διαφορά. Δεν είναι κυδανικό. Ευχαριστώ συνάδελφοι για την υπομονή σας. colleagues, um, my apologies. Ζητώ συγγνώμη, συνάδελφοι. Θα έπρεπε να αρχίσει ε, το επόμενο θέμα. Καθίστε, πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε. We are very much, um... Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Παρακαλώ, ε, καθίστε. Να ξέρω ότι καθυστερήσαμε να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες, αλλά καθίστε. Έχουμε την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης ε, του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Ξέρω ότι ήταν μακρά η ψηφοφορία. Καθίστε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Παρακαλώ και τους ε, υψηλόβαθμους υπαλλήλους εκεί πίσω και τους συναδέλφους που είναι όρθιοι να καθίσουν. Λοιπόν, έχουμε την έκθεση το 2014 για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σήμερα έχουμε προσκαλέσει την κυρία Φράουκε Ζάιτενστίκερ, Γνωριζόμαστε, ξέρετε ότι με την προφορά δεν τα πάω καλά, που είναι η νέα πρόεδρος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από το Μάρτιο του 2015. Έχουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Μανολόπουλο, που είναι μεταβατικός ε, διευθυντής. Ε, Σας καλωσορίζω θερμά. Πολύ σημαντική δουλειά κάνατε τη μεταβατική αυτή περίοδο για την κοινή συζήτηση. Έχουμε επίσης παρόντα εδώ ενώπιόν μας ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο εξίσου. VIP είναι και ο κύριος Πολ Νέμιτς που ήταν και χτες στο τριμερή διάλογο για τον κανονισμό. Και πολύ καλός φίλος και παλιός γνώριμος, διευθυντής για τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης Justice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλωσορίζω λοιπόν όλο το πάνελ. I'm to start, I think, with, um... Αρχίζουμε. Ο Παουλ Νέμιτς. Ποιος θα αρχίσει πρώτος. Α. Αυτά γίνονται μετά από μεγάλες και μακρές ψηφοφορίες. Θα ακούσουμε πρώτα λοιπόν την κυρία Ζάιτεν Στίκερ και μετά τον κύριο Μανολόπουλο και μόνο στη συνέχεια τον Πολ Νέμιτς που θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων με αυτή τη σειρά. Λοιπόν, η κυρία Ζάιτεν Στίκερ πρώτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το μικρόφωνο δουλεύει μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καλημέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας. Μια στιγμή, συνάδελφοι, παρακαλώ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι ενώπιον σας για να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση του οργανισμού μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σας, ειδικά τα μέλη της Επιτροπής σας, για τις προσπάθειες που κάνετε ε, να μπουν τα θεμελιώδη δικαιώματα σε τόσους τομείς πολιτικής, όπως είδαμε σήμερα. Οι σημερινές συζητήσεις ελπίζω να σας υποστηρίξουν για τις απερχόμενες συζητήσεις για την έκθεση του Κοινοβουλίου ως προς την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν καλύψει ο κύριος Μανολόπουλος κάποια βασικά σημεία που μας ανησυχούν, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τις αλλαγές που κάναμε και στη δομή αλλά και ε, στην έκταση της σημερινής και φετινής έκθεσης στο παρελθόν ήταν ένας κατάλογος 300 σελίδων, μια απογραφή των εξελίξεων στα θεμελιώδη δικαιώματα. Εμείς το έχουμε περιορίσει και έχουμε επιλέξει τομείς στους οποίους μπαίνουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Στα τέλη του περασμένου έτους ε, ήταν η πέμπτη επέτειος από τη συνθήκη της Λισαβόνας, που σημαίνει ότι ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει πενταετή ήδη εφαρμογή και έχει έρθει η ώρα να, αξιοποιήσουμε, να αξιολογήσουμε μάλλον τα υπέρ και τα κατά και τις αδυναμίες τους. Γι' αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της φετινής ε, έκθεσης είναι αφιερωμένο στο χάρτη και στις επιδόσεις των 28 κρατών μελών. Αυτό επιτρέπει εξέταση του ρόλου του χάρτη ε, εθνικά δικαστήρια. Πράγμα που είναι πάρα πολύ εύγλωτο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τους Ευρωπαίους πολίτες τέτοια θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στην καθημερινή του ζωή. Προχωρώντας θα ήθελα να μπω σε κάποιες λεπτομέρειες ως προς την εστίαση που είναι το προήμιο όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Πέρυσι είχαμε ασχοληθεί με ένα στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, αναζωογονηθεί ε, η ε, προσήλωση της νεολαίας στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και φέτος έχουμε αφοσιωθεί στους δείκτες. Τι στόχο έχουν και ποια είναι η λειτουργία τους. Η μία λειτουργία τους είναι να βελτιώνεται η συγκρισιμότητα και η αντικειμενικότητα των στοιχείων και των δεδομένων. Αν γνωρίζουμε περισσότερα για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη, θα είναι και καλύτερο ο πλήρη σεβασμό τους. Για να ταυτοποιούμε λοιπόν, να συλλέγουμε και να αναλύουμε αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει οι δείκτες να αντανακλούν το τι κάνουν τα κράτη-μέλη και τι αποτελέσματα έχουν όλα αυτά. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ένα πλαίσιο που θα ενταχθούν. Είπα ότι αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει εκπονήσει δείκτες ε, που είναι πάρα πολύ κατάλληλοι και μετρούν και τα αποτελέσματα αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται για να φτάνουμε σε αυτά. Και ο δικός μας οργανισμός χρησιμοποιούμε το ίδιο ε, εργαλείο και έχουμε τρεις κατηγορίες δικτών. Έχουμε διαρθρωτικούς, διαδικαστικούς και ε, δείκτες που μετρούν το αποτέλεσμα εξετάζουν πρώτα το νομικό πλαίσιο, το σύστημα εφαρμογής και την πραγματική κατάσταση επιτόπου. Το 2007, απαντώντας σε αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οργανισμός μας άρχισε να εκπονεί ένα τέτοιο πλαίσιο για δείκτες για να ε, συλλέγουμε και να αναλύουμε στοιχεία για τα δικαιώματα των παιδιών ακολούθησε ένα πλαίσιο δικτών για τομείς ε, δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία και για Ρωμά. 17 κράτη-μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει για ένα κοινό πλαίσιο παρακολούθησης της ένταξης ε, που έχουμε εκπονήσει στην ομάδα εργασίας μας για τους δείκτες ε, ως προς τους Ρωμά. Βέβαια, όποιο τομέα και αν έχουν σχεδιαστεί να μετρούν αυτοί οι δείκτες, έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι καλά σχεδιασμένοι και να στέκουν πάρα πολύ από επιστημονικής πλευράς. Και θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και οι ε, ελεγχόμενοι, να βασίζονται σε παραμέτρους και μεθοδολογικά κριτήρια. Επίσης, να υπάρχει μια σαφής κανονιστική ερμηνεία και να ε, χρησιμοποιούνται γρήγορα και άμεσα τα δεδομένα και τα στοιχεία. Έτσι θα μετρούμε όχι μόνο το αποτέλεσμα αλλά και τις προσπάθειες να βελτιωθούν ε, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και να αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις. Έτσι θα μπορέσει να ενταχθεί παντού αυτή η υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Ε, έτσι θα ενισχυθεί και η λογοδοσία και η διαφάνεια των αρχών και σε ευρωπαϊκό και σε κρατικό επίπεδο, μιλώντας πάντα στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί αυξάνεται η καχυποψία και η δυσπιστία, όχι απέναντι μόνο σε πολιτικούς, αλλά σε θεσμούς και θεσμικά όργανα ολόκληρα. Αυτά τα μέτρα δεν μπορούν παρά να ενισχύσουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Θα ήθελα τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μανολόπουλο για να πει σε περισσότερες λεπτομέρειες για κάποια βασικά θεμελιώδη δικαιώματα και προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στην ετήσια έκθεσή μας φέτος. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από πλευρά μου για την πρόσκληση που λάβαμε για να σας παρουσιάσει ο οργανισμός μας την ετήσια έκθεση για τις προκλήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, αναφέρθηκε, εξορθολογίστηκε η έκθεση φέτος για να έχουμε μια πιο στοχευμένη ανάλυση. Η έκθεση καλύπτει τους τομείς ε, που καθορίζονται από το ετήσιο πλαίσιο που καθορίζει τους τομείς ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων στους οποίους ε, ε, κάνει επεξεργασία ο οργανισμός μας για πέντε χρόνια. Έχουμε διακρίσεις, ένταξη των Ρωμά, άσυλο, θεωρήσεις, μετανάστευση, κοινωνία της πληροφορίας, προστασία δεδομένων, δικαιώματα του παιδιού και πρόσβαση σε δίκη, ακόμα και τα δικαιώματα των θυμάτων. Επίσης στην έκθεση θα βρείτε και ένα κεφάλαιο για την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη χρήση τη στα κράτη-μέλη. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε για όλη την έκθεση. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία θέματα όμω, ε, για τα οποία έχουμε αρκετά αποτελέσματα στην έκθεση και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το 2014 και για το 2015. Τη μετανάστευση, τα δικαιώματα των θυμάτων και τα δικαιώματα του παιδιού. Σήμερα το πρωί έγινε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για τη μετανάστευση και με εξέπληξε ε, αυτό το οποίο είπε ο δημοσιογράφος που χρησιμοποιούν κάλυψη για να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι κάνουν και μετανάστευση ε, αυτό το οποίο συζητούμε. Να Πλησιάζω λοιπόν στη μετανάστευση και το άσυλο. Πρόκειται για θέματα τα οποία παραμένουν επίκαιρα στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο και όπως γνωρίζετε οι τραγωδίες στο Μεσόγειο, στη Μεσόγειο επιδεινώθηκαν. Ε, είχαμε θάνατο ακόμα περισσότερων ανθρώπων στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη. Ε, φέτος ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ ψηρότερος, όπως εκτιμά ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης διότι πάνω από 800 άτομα πέθαναν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου. Ε, γνωρίζουμε άλλωστε και τα γεγονότα στη Λαμπεντούζα. Αυτός ο τραχικός χαμός ανθρώπων πρέπει να σταματήσει και γι' αυτό και ακριβώς ε, ε, χαιρετίζουμε και την έκθεσή σας για την ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης για τη μετανάστευση. Ο οργανισμός μας προσφάτως δημοσίευσε και μία έκθεση με ε, αρκετά επιχειρήματα ε, και υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες όχι μόνο βοηθούν να σωθούν ζωής αλλά βοηθούν και στην καταπολέμηση της εμπορίας ε, ανθρώπων και της διακίνησης ανθρώπων. Υπάρχουν δύο βασικές προκλήσεις για το άσυλο. Καταρχάς υπήρξε επιδίνωση στα σύνορα των κρατών μελών όσον αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης. Ε, κανείς δεν θα πρέπει να επαναπροωθείται σε μια χώρα στην οποία η ζωή του ή η ελευθερία του είναι σε κίνδυνο. Δεύτερον, δύο χρόνια μετά τη την λήξη της ε, ημερομηνία μεταφοράς, ακόμα δεν υπάρχει σε κάποια κράτη-μέλη ένα σύστημα παρακολούθησης για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συμμόρφωση για τις αιτήσει ασύλου και για τις διαδικασίες επιστροφής των ατόμων ε, που ε, έχουν απορριφθεί αιτήσει. Υπάρχουν ε, ε, στοιχεία και που καταδεικνύουν επίσης ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία στους, ε, στα τμήματα τα οποία είναι υπεύθυνα για τις επιστροφές. Πολλές φορές οι μετανάστες είναι θύματα διάκρισης, εγκριμάτων μίσους και πολλά κράτη-μέλη έχουν κάποιες πολιτικές και μέτρα για να το καταπολεμήσουν, αλλά η εφαρμογή υστερεί και υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι υπάρχουν, παρακολούθηση, υπάρχει παρακολούθηση και έλεγχος για τις συνέπειες. Πολλές ε, ε, είναι οι λύσεις. Παραδείγματος χάρη, το 2014 12 κράτη-μέλη ε, εφήρμοσαν ε, προγράμματα κατάρτισης ε, για προσωπικό το οποίο ασχολείται απευθείας με μετανάστες και είδαμε ολένα και μεγαλύτερο αριθμό χωρών να αναγνωρίζει ότι η ένταξη δεν αφορά μόνο τους μετανάστες και τα παιδιά τους, αλλά όλη την τοπική κοινότητα. Αυτό από μόνο του βέβαια δεν βελτιώνει και πάρα πολύ τα ποσοστά επιτυχίας ένταξης των μεταναστών. Τώρα να σταθώ λίγο στο θέμα των θυμάτων εγκλήματος. η έρευνα μετά από την εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων ε, καταδεικνύει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν περισσότερα μέτρα για να διασφαλίσουν ε, κατάλληλη προστασία. Καταρχάς, ε, δικαίωμα στην ενημέρωση των θυμάτων φαίνεται ότι είναι πρόβλημα σε αρκετές χώρες. Εδώ δεν πρόκειται απλώ για νομική συνδρομή, αλλά και για ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη, κάτι το οποίο θα πρέπει να παράσχεται στα θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις διάφορες ποινικέ διαδικασίες. Στα περισσότερα κράτη-μέλη ε, πρέπει να έχει γίνει μεταφορά της οδηγίας για τα θύματα και ακόμα υπάρχει καθυστέρηση και κρεμούν πολλά. Έγινε μια συνάντηση με τον Επίτροπο και 8 κράτη-μέλη στη Βιέννη την προηγούμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε την εφαρμογή και τη μεταφορά της οδηγίας για τα θύματα και νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά υπάρχουν και παραδείγματα που είναι καλά. Παραδείγματο χάρη, σε αρκετά κράτη-μέλη συλλέγονται χρήματα για στήριξη των θυμάτων μέσω ενό ταμείου, στο οποίο ε, καταβάλουν ποσά. Ε, για τα θύματα. Παραδείγματο χάρη, η Φιλανδία έχει χρέωση 8 ευρώ για άτομα που έχουν διαπράξει κάποια εγκλήματα και τα χρήματα πηγαίνουν σε υπηρεσίε στήριξη των θυμάτων. Το ταμείο αυτό αναμένεται να ε, συλλέγει ένα σημαντικό ποσό κάθε χρόνο και καλούμε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν και άλλα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να έχουμε πλήρη υποστήριξη προς τα θύματα και να υπάρχει πρόσβαση στα μέτρα αυτά από τα θύματα. Πρέπει για παράδειγμα να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, να διασφαλίσουμε δίκαιη δίκη και να υπάρχει και επιμόρφωση αστυνομικών και άλλων ε, υπαλλήλων για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν ε, τους ανθρώπους αυτούς στη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τα θύματα δεν θα καταγγέλουν τις εμπειρίες τους και χωρίς κατάλληλες καταγγελίες δεν μπορούμε να διώξουμε τους δράστες ή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού το 1 τρίτο των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Και ο κίνδυνο αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό σε κάποιε χώρε. Οι οικογένειε με παιδιά δυσκολεύονται να πληρώσουν τα δάνειά του, τη θέρμανση, το σχολικό υλικό ε, και ακόμα και βασικά τρόφιμα. Επομένως πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια των παιδιών και να συμπεριληφθούν αυτά στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Νομίζω ότι ο πρόεδρος αναφέρθηκε στους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο ή πρόεδρος παιδιά θύματα βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης ή άτομα χωρίς κυδαιμονία, παιδιά χωρίς γονείς ή κυδαιμόνες. Ε, ε, είναι θέματα τα οποία μελετήσαμε, αλλά δυστυχώς ε, διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα δεν επαρκούν και δεν υπάρχουν και κατάλληλοι πόροι για να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρέ οι προκλήσει στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα στη ε, θέματα μεταχείριση και συμπεριφορά προ τα παιδιά σε ποινικέ διαδικασίε, ε, ε, σε συνεργασία με δικαστέ, δικαστικό προσωπικό, ε, αστυνομικούς ε, και λοιπούς. Κυρίες και κύριοι, θα έπρεπε να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα χώρο ελευθερίας και ασφάλειας για τους πολίτες της. Έχουν γίνει πάρα πολλά ε, και το πλαίσιο θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι συμπαγές, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα, γι' αυτό και ακριβώς η συνεργασία μαζί σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστούμε. Δεν ε, ήθελα ε, να φύγουν όλα τα μέλη της Επιτροπής, ε, ήθελα να γίνει εγκαίρως η παρουσίαση και εγώ πρέπει να φύγω στις 12 και 20 και διάφορα άλλοι μέλη της Επιτροπής θα φύγουν και δεν θέλω να χάσουμε τις ερωτήσεις και γι' αυτό σας πίεσα. Θέλεις τώρα να μιλήσεις πριν να αρχίσεις γιατί θα φύγω 12 και 4. Ε, και πρέπει να μας πούν ε, ε, και οι συνάδελφοι, θα, θα σας ακούσουμε όλους, σε κάποιος θα με αντικαταστήσει. Απλώς ήθελα να σας ευχαριστήσω ήδη τώρα γιατί μπορεί να έχω φύγει. κάτι που απασχολεί τα μέλη της Επιτροπής μας, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας, είναι ότι προς το παρόν έχουμε τρεις μηχανισμούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με το διάλογο που έχουν ε, σε σχέση με τις παρεμβάσεις ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα διότι υπάρχουν παραβιάσεις από πλευράς κρατών μελών πλέον συχνά και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει αυτό για πολύ βασικά ζητήματα και ένας τομέας είναι ο δικός σας τομέας δράσης. Έχουμε το άρθρο 2 το άρθρο 7, ξέρουν όλοι πόσο ε, εκμηρό εργαλείο είναι αυτό. Για το Κοινοβούλιο όμως είναι περίπλοκη η κατάσταση, διότι αμφισβητούμε το πότε, το πώς παρεμβαίνουμε ακόμη και τους μηχανισμούς, τα δικαιώματα του Προέδρου, τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Όλα αυτά πέφτουν πάνω στην Επιτροπή μας. Εσεί είστε από την Επιτροπή και είναι παράδειγμα να σας ρωτώ ε, για το ρόλο του Κοινοβουλίου, αλλά είναι ένας τομέας που έχει μια δυναμική και κάνουμε τη δουλειά μας, θέλουμε να την κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Πώς, πώς όμως πρέπει να την κάνουμε και αυτό είναι το ζήτημα που μας απασχολεί. Είναι συναρπαστικό αυτό ο τομέα και πολύ σημαντικό το ζήτημα. Αν μπορείτε να μα δώσετε τα φώτα σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια και μετά θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις στις συγκεκριμένες ερωτήσεις του Πρόεδρου. Ο πρόεδρο Γιούνκερ έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων που έχει ε, στον τομέα των αρμοδιοτήτων τη και να Διαφυλάται και να προωθεί τις βασικές μας αξίες. Ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαν στην Επιτροπή, είπε, στην Επιτροπή σας είπε ότι εάν θέτουμε κινδύνο τις αξίες μας, θέτουμε κινδύνο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την ετήσια έκθεση για την ε, υλοποίηση της Χάρτας των Μελωδίων Δικαιωμάτων προκύπτει από τον ε, Οδικό Χάρτη του 2010 για την εφαρμογή ε, του χάρτη, εργαλείο παρακολούθησης δηλαδή των προκλήσεων όπου εκλήθη να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνοντας πώς λήφθη υπόψη ο χάρτης στην νομοθετική διαδικασία, στην εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων από εκτελεστικά όργανα καθώς και στην ομολογία. Ας αρχίσω από το τελευταίο, την ομολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαστήριό της χρησιμοποιεί ένα και περισσότερο τη σύμβαση ε, παρατίθεται ε, τμήματα της σύμβασης. Ε, το 2014 210 φορές αναφέρθηκε το δικαστήριο στη, στη χάρτα σε σχέση με 114 φορές το 2013, 97 το 2013 και 43 το 2012. Ζει και βασιλεύει ο χάρτης ε, στην ομολογία και απεδείχθη αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τα κράτη-μέλη. Ε, για την κατάργηση της απόφασης ε, της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας. Είχαμε πολύ μια σημαντική απόφαση. Επίσης είχαμε την απόφαση ΣΕΚΕΡ για τα, τη Γεωργία την Αλία, όπου επίσης αναφέρθηκαν τα δικαιώματα και βλέπουμε ότι ε, πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση από τα τρία θεσμικά όργανα, συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους για διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τόσο ώστε μετά να μην ε, προσβάλλονται, να μην ε, γίνονται προσφυγές εναντίον τους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχει διαδικασία streamlining ε, καθ' όλη τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου από την κατάρτιση των προτάσεων μέχρι την έγκριση και την υλοποίησή τους. Ε, το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα της πολιτικής. Αυτό κάνουμε εμείς στην υπηρεσία μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα άλλα θεσμικά όργανα για τις τροπολογίες, τις ουσιαστικές, abstantive τις ουσιαστικές τροπολογίες που καταθέτουν. Ε, τα, συστηματικά πρέπει να γίνεται αποτίμηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα καθ' όλη τη ε, διάρκεια του νομοθετικού κύκλου και την βάση του πακέτου για την καλύτερη νομοθετική διαδικασία υπάρχει πρόβλεψη συστηματικά να γίνεται αξιολόγηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα έχουμε τη νέα διαθεσμική συμφωνία. Ε, η οποία ελπίζουμε θα λειτουργήσει ως πλαίσιο για να συζητούμε τον τρόπο με τον οποίο και οι συνομοθέτες μπορούν να ενισχύσουν την αποτίμηση που κάνουν για την ε, ε, τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον έλεγχο που κάνουν των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2014 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη για την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το πώς πρέπει να κινηθούμε. Η προσχώρηση παραμένει προτεραιότητα και έτσι αυξάνεται η προστασία των θεμελιδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτω χρονική στιγμή τη προσχώρηση, εάν υπογραφεί συμφωνία, τόσο άλλου χρειάζονται χρόνια, διότι πρέπει μια τέτοια συμφωνία να επικυρωθεί από όλα τα συμβαλώμενα μέρη. Όσο χρόνο και αν πάρει, φέρουμε την υποχρέωση να λάβουμε δέοντος υπόψη την ομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις πρακτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα η παρακολούθηση της εφαρμογής του χάρτη κατά την εφαρμογή του νοσιακού δικαίου και αυτό είναι ένα τμήμα της ετήσιας έκθεσης. Ε, και τώρα φτάνω ε, στο πρώτο εργαλείο που έχουμε το 2014 ξεκίνησαν 11 διαδικασίε επί παραβάση κατά κρατών μελών ε, με στόχο να μεριμνήσουμε ούτω ώστε να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του χάρτη. Και επανέρχομαι στην ερώτησή σα, Πρόεδρε, για να είμαι πολύ συγκεκριμένο, Ήδη αναφέρθηκα σε δύο βασικού τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρεμβαίνουν Είναι κέρια σημασία. Πρώτον, στην νομοθετική διαδικασία, σε επί, ε, διακεκριμένη ακαδημαϊκή έδειξαν ότι από τότε που άρχισε να έχει νομοθετικέ αρμοδιότητες ε, το Ευρωπαϊκό το επίπεδο διαφύλαξη των δικαιωμάτων σε τομεί πολιτική ε, αυξάνεται διαρκώ από τότε που συναποφασίζει το Κοινοβούλιο. Βλέπετε λοιπόν με την παρέμβαση του Κοινοβουλίου προστατεύονται καλύτερα τα μεμονωμένα δικαιώματα και εμπειρικά έχουμε διαπιστώσει πω η προκάτοχη σα και εσεί ε, το έχετε κάνει. Δεύτερον, έλεγχο τη εκτελεστική εξουσία με δύο τρόπου. Πρώτον, έλεγχο Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να υπάρχει σωστή ε, άσκηση των αρμοδιοτήτων μας και αναφέρθηκε σε 11 διαδικασίες επί παρέμβαση και θα φτάσω και στο μηχανισμό του άρθρου 7 που αναφέρεται αλλά και έλεγχος της εκτέλεσης ε, του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι αυτή είναι φυσική λειτουργία του Κοινοβουλίου, δηλαδή κοιτάζει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων στους ώστε να υπάρχει σωστή εφαρμογή της χάρτας Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ καλό να εξετάσουμε μονομένες περιπτώσεις το Κοινοβούλιο, στα κράτη-μέλη δηλαδή, που ε, φέρουν επίσης υποχρεώσεις ε, σωστής εφαρμογής ε, του νόμου. Πού έχουμε ανησυχίες για τις διαδικασίες παράληψης. Άσυλο και μετανάστευση φυσικά σε σχέση ε, με την ε, έλλειψη ενδίκων μέσων, συνθήκες εκράτησης, ε, συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και το καθεξής. Για το 2014 με πρόταση αναθεώρηση του Δουβλίνου 3 για την εξέταση αιτήσεων ασύλου από ασυνόδευτούς ανήλικους προτείνουμε να ληφθεί υπόψη η νομολογία του δικαστηρίου ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα των παιδιών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω πόση σημασία αποδίδουν δούμε στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη ένα οριζόντιο δικαίωμα που κατοχυρώνεται για όλους. Είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Το 2014 ε, απευθύναμε όκληση προς τα πέντε κράτη-μέλη σε σχέση με αποφάσεις ανάκλησης ή ε, κατάργησης ε, θεώρησης χωρίς πρώτερη προσφυγή σε δικαστικό όργανο. Επίσης, ε, ε, υπάρχουμε το πακέτο των οικονομικών μέτρων ε, Παραδείγματο χάρη, ε, ρήτρε διαφύληξη, ε, τεκμήριο αθωότητας και νομική συνδρομή για τα παιδιά. Όταν εγκριθεί αυτό το πακέτο θα ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και έτσι θα αρχίσει να λειτουργεί πιο εύρυθμα η αμοιβαία αναγνώριση στου δικονομικού κανόνε και θα ενισχυθούν τα παιδιά σε ποινικέ διαδικασίε. Θα ήθελα να σας επιθυμήσω και πάλι ότι στα πλαίσια του ψηφιακού περιβάλλοντος υιοθετήθηκαν οι κανόνε για την προστασία. Αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία Τέλο του τρέχοντος και νομίζω είναι προτεραιότητα όχι μόνο για την Επιτροπή αλλά και για το Κοινοβούλιο. Αν να μην ξεχάσω, να σας παραπέμψω και στο ειδικό τμήμα Focus μέσα στην ετήσια έκθεση για το χάρτη που σχετίζεται με την ψηφιακή κοινωνία, τα μεγάλα δεδομένα Big Data τα ογκώδη μάλλον δεδομένα και οι, μεγάλοι, οι νέες ε, δυνατότητες που πρέπει να συνοδεύονται από μεγάλη εμπιστοσύνη και στην προστασία των δικαιωμάτων για τα εγκλήματα μίσου και τον αντισημιτισμό και, και την Ισλαμοφοβία. Ε, έχουμε πρόσφατα ανησυχητικά φαινόμενα, αλλά όπως και την, σε σχέση με την ομοφοβία, την αφροφοβία, ε, έχουμε απαράδεικτα φαινόμενα που και βλέπουμε ότι έχουμε, ε, έχουν σημειωθεί και πολλά περιστατικά ε, βίας. Ε, ο, ο αντιπρόεδρος Τίμερμαν ε, την 1η και 2 Οκτωβρίου 2015 θα μιλήσει συγκεκριμένα για την ανεξιθρησκεία, κυρίως για την καταπολέμηση του μίσους κατά των οπαδών του Ισλάμ στην Ευρώπη. Από το 2008 και μετά υπάρχει και το θέμα της οδηγίας για να καλυφθούν τα χάσματα. Ναι, ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και έχουμε μόνο 15 λεπτά. Θα φύγω κι εγώ και θα μείνετε μόνο σας εδώ. Και θα είναι πραγματικά ψηφιακά τα δικαιώματα γιατί θα είναι εικονικά, δεν θα έχετε κανένα να τα πείτε. Ε, λοιπόν, έχουμε και την συνεδρίαση με το Συμβούλιο και πρέπει να πάω και ο Πίτερ παρακαλείται να έρθει εδώ να αναλάβει την Προεδρία. Ε, για τη σύγχυση ανάμεσα στο άρθρο, με το άρθρο 2, μπορείτε να μας μιλήσετε, έχετε όλους τους αγωνιστές εδώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι συνάδελφοι λοιπόν χρειάζονται μια σαφή απάντηση. Πώς παρεμβαίνει το Κοινοβούλιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Γίνονται περίπλοκα τα πράγματα διότι έχουμε ε, τη δική σας υπηρεσία αλλά έχουμε και εμείς ένα ρόλο και θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας αλλά περιπλέκονται τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να το θέσω και πάλι. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, μας βοηθήσει σε σχέση με την ε, δράση που έχουμε στα κράτη-μέλη, σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής ε, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντες για μας. Θέλουμε σαφήνεια με ποιο τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε. Επίσης η διαδικασία του διαλόγου και εκεί επικρατεί ασάφεια. Ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο του διαλόγου. Θα ήθελα να διευκρινιστούν αυτά. Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συμβάλλουμε σε αυτό που εσείς πετύχατε και που βλέπουμε στην ετήσια έκθεση. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά αν μπορείτε να εστιάσετε σε αυτό το σημείο. Okay, thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε μερικούς ομιλητές. Η ε, πρώτη είναι η Μαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους ε, τους ομιλητές και για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό, το είπε και ο Κλοντ, να έχουμε την συνολική εικόνα, την αντικειμενική και με συγκρίσιμους δείκτες. Ε, αν έχουν ανταποκριθεί ε, τα κράτη-μέλη στι υποχρεώσει τους ή όχι ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και πρώτη ερώτηση προς τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Λέω ότι είναι κάπως σκληρό αυτό, αλλά Τώρα με αυτό το σύστημα δικτών που έχετε εσείς υιοθετήσει, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκριτική αξιολόγηση και εκτίμηση του τρόπου εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων για να υπάρχει αναφορά. Πολύ ωραίο είναι να μας δίνετε τους δείκτες, αλλά είναι μισή δουλειά. Και ένα δεύτερο, θέλω να σας συγχαρώ για την κοινωνία των πολιτών και το σχετικό κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να ρωτήσω τον Πάουλ Νέμιτς και άλλους που ασχολούνται με αυτό. Για την προστασία των δεδομένων. Τι γίνεται με θέμα παρακολουθήσεων και μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι 12 κράτη-μέλη ε, αδυνατούν απολύτως να προστατεύουν τους πολίτες τους κατά παρακολουθήσεων, υποκλοπών κτλ. Ιδιωτική ζωή, προστασία που παραβιάζονται από τις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή αυτό που συζητούμε εξαιρεί αυτές τις υπηρεσίες από την παρακολούθηση και τις προστασίες των δεδομένων. Ακούω τις συστάσεις ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά αυτά πώς τα εφαρμόζετε και τι κάνετε για αυτό. Και τι γίνεται με τις άλλες υπηρεσίες, τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών, διότι δεν ε, προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δεδομένα, τα προσωπικά. Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις, θα τις ομαδοποιήσουμε. κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε και οι δύο εκθέσεις που συζητούμε σήμερα αφορούν το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και πώς εφαρμόζεται, και μάλιστα πώς εφαρμόστηκε το 2014. Φαίνεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου όμως, διότι δεν ασχολούνται καθόλου με το σημαντικότερο θέμα ε, παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η δολοφονικές πολιτικές λιτότητες που πλήττουν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και απορρέουν ε, από τα θεσμικά όργανα. Ούτε καν αναφέρονται ούτε στην έκθεση της ΦΡΑ ούτε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή υπονοείται πραγματικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μη εφαρμογή των κοινωνικών και ε, οικονομικών δικαιωμάτων ή απλώς υποδίεστε ότι δεν υπάρχουν ή τα ξεχνάτε. Το κεφάλαιο 4 στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει τον τίτλο Αλληλεγγύη και προβλέπει μεταξύ άλλων το δικαίωμα στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις, άρθρο 28, το δικαίωμα στην προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, το άρθρο 30, δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, άρθρο 34 και δικαίωμα στην ε, γενομική περίθελψη άρθρο 35. Όλα αυτά τα άρθρα παραβιάζονται από πολιτικές που επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στα κράτη-μέλη της Ένωσης, π.χ. στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως μέλη της Τρόικα έχουν ακυρώσει τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις, περικόψει μισθούς και συντάξεις ε, σε ε, χαμηλότερο βαθμό από το ελάχιστο επιβίωσης. Έχει αυξηθεί η θνησιμότητα ε, γύρω στο 15% κτλ. Πολλά από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά τις απαιτήσεις της Τρόικα ε, αποδεικνύονται ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων μέσω αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και παραβιάζουν και πολλές συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας μετά από αποφάσεις του ILO. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι προφανές ότι όταν υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις τέτοιων μέσων διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αντίστοιχα παραβιάζονται και άρθρα και δικαιώματα που εγγράφονται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Παρόλα αυτά, τα εν λόγω θεσμικά όργανα όχι μόνο δείχνουν απροθυμία να συμμορφωθούν με αυτά τα ευρήματα, αλλά απαιτούν από τη νέα ελληνική κυβέρνηση μέσα στο πλαίσιο των συνεχιζομένων διαπραγματεύσεων για το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής και άλλες παραβιάσεις κοινωνικών δικαιωμάτων εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών και αυτό είναι ένα μόνο τμήμα του γενικότερου προβλήματος παραβιάσεων κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου, αλλά και γενικότερα σε πολλά κράτη-μέλη, μέσω των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται. Ε, είναι σχεδόν σαν να ζούμε σε, σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα ε, ως προς την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιδών Δικαιωμάτων και σήμερα και το 2014, στο οποίο αναφέρεται η εκθέσή σας και οι δύο εκθέσεις. Και νομίζω ότι είναι έσχος το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνονται. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, επομένως θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε λίγο πιο λακωνικοί στις παρεμβάσεις σας, αν γίνεται. Η κυρία Ντελάζ. Ευχαριστώ. Θα περάσω απευθείας σε ερωτήσεις μου. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας. Πρώτη μου ερώτηση προς την υπηρεσία. Για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αριθμός των προσφύγων ε, των, ε, του άσυλο έχει υπερβεί τα, τα 50 εκατομμύρια, ε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Επειδή οι δυνατότητε ε, εισόδου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περιορισμένε, και τα άτομα τα οποία χρειάζονται προστασία εξακολουθούν να μην έχουν λύσει. Τι εκτίμηση κάνει η υπηρεσία για τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως για τους νόμιμους διάβλους μετανάστευσης και για τους λεγόμενους οικονομικούς μετανάστες. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις στρατηγικές μας στα συγκεκριμένα σημεία. Μία ερώτηση προ την Επιτροπή τώρα. Στο τελευταίο τμήμα τη έκθεση σα για την εφαρμογή τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη ψηφιακή στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει την υποχρέωση το ε, ύπαρξη διαδικτυακή πλατφόρμα για θέματα τρομοκρατία, οργανωμένου εγκλήματος και καταπολέμησής του. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας αυτή τη πλατφόρμα με τι αρμόδιε αρχέ για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και τα μηνύματα μίσου ε, στο διαδίκτυο. Σε ποιο βαθμό ε, θα πρέπει να γίνεται αυτή η συνεργασία. Μπορούμε να έχουμε και πιθανές κυρώσεις ε, κατά ε, όλων αυτών που θα αρνηθούν στο διαδίκτυο να συνεργαστούν. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς ε, την ε, παρουσίαση για τον έλεγχο που έχει διεξαχθεί και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον υπάρχει η ίδια προσοχή και παρακολούθηση για τα ίδια τα θεσμικά όργανα και το πώς ε, τηρούν αυτή την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και με ποια κριτήρια. Και πώς θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κρίνει τη συμπεριφορά του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, το ερώτημά μου αφορά δύο τομείς. Καταρχάς την πολιτική μετανάστευση, το κοινοτικό σκέλος της πολιτικής μετανάστευσης και πιο συγκεκριμένα πολιτικές όπως ε, το θεματολόγιο της μετανάστευσης το οποίο συζητάτε αυτές τις μέρες. Βρισκόμαστε ενώπιον πολύ σοβαρών κινδύνων παραβίασης της χάρτας, ιδίως ε, το θέμα της μη επιστροφής, της μη επαναπροώθησης και επίσης σε κοινοτικό επίπεδο υπάρχουν κάποιες προτάσεις για νόμιμους διάβλους ε, διαφυγής από χώρες ε, που βρίσκονται σε κατάσταση σύρεξης, όπως εσείς αναφέρετε, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν αναφέρεστε σε αυτό για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα στα κράτη-μέλη ή για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται σεβαστά από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Και δεύτερον, θα ήθελα να συμπληρώσω ε, στα όσα είπε ο συνάδελφο Χρυσόγονο. Οι πολιτικέ λιτότητε ε, και οι συνέπειε στα θεμελιώδη και κοινωνικά δικαιώματα. Βρισκόμαστε ενώπιον ε, μια συστηματικής παραβίασης της χάρτας και των ίδιων των συνθήκων. Η λιτότητα είναι από μόνη της συστηματική παραβίαση των συνθήκων και δημιουργεί μια πολύ επικίνδυνη απόκληση μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών και ε, λαϊκής ετοιμογορίας ε, και αποτελεσμάτων των εκλογικών αναμετρήσεων. Θα πρέπει κάπου όλα αυτά να τα σταθμίσουμε και να ε, δούμε τι ισχύει. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι πολλές παραβιάσεις, τις οποίες αναφέρεστε εσείς πολύ σωστά στην εκθεσή σας, ε, εγκλήματα μίσους, ξενοφοβία, Ε, άρνηση της διαφορετικότητας, η Ισλαμοφοβία σχετίζονται με ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες σε κοινοτικό επίπεδο παραβιάζουν τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ε, ως αντίδραση έχουμε μεγάλα κύματα ξενοφοβίας ε, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες είναι η τελευταία μελήτρια. Σας ευχαριστώ για την έκθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως για τα σχόλια που κάνατε, για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα θέματα της μετανάστευσης και της αρρωγής προς τους ε, τούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Α, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλες σημαντικές προφορές μέσα στην έκθεση. Πιστεύω όμως ότι όντω πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο, μια αναχώρα έκθεση για, για τις 28, για να έχουμε πληρέστερη εικόνα. Διότι Αυτά που μας είπε ο κύριος Χρυσόγονος και η κυρία Σπνέλη μας είπαν τώρα θα τα αναφέρονταν μέσα στην έκθεση άμα είχαμε αναχώρα ε, κεφάλαιο. Δηλαδή το φοβερό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι πολιτικές στις χώρες, ε, οι πολιτικές της Τρόικα παραδείγματος χάρη, ε, όπου βλέπουμε τις ε, συγκεκριμένες ευθύνες που έχουν και η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ισχύει και για τη χώρα μου. Το λέτε εσείς, λέτε ότι στη χώρα μου, στην Πορτογαλία, ότι τα παιδιά ε, με κίνδυνο φτώχειας ε, πλέον έχουν ξεπεράσει το 1 τρίτο των παιδιών της χώρας. Είναι φοβερός αυτός ο δείκτης ε, σε σχέση με την επιδείνωση της κατάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να επιδεινώνεται διότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για χαμένες γενιές. Ε, για να μην αναφερθώ στους ανέργους νέους που επίσης ε, είναι μια άλλη χαμένη γενιά και όλες τι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο οποίο αυτό μας οδηγεί γιατί υπάρχει ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού πέρα από τους πλέον ευάλωτου, όπως ε, η ΡΟΜ, όπως ε, η, η ΑΜΕΑ και σε χώρες όπως η Πορτογαλία και το ξέρω ότι και στην Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει και στην Ιρλανδία είναι ανίποτα τα βάσανα που υπομένουν αυτοί οι άνθρωποι γιατί υπάρχει και το δικαίωμα στη ζωή πολλοί ε, έχουν αυτοκτονήσει και ξέρω γιατί μιλάω, ξέρω ε, συγκεκριμένα περιστατικά στην Πορτογαλία. Λοιπόν, θα έλεγα πως χρειαζόμαστε έκθεση αναχώρα, ούτω ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η παρακολούθηση μέσω της ετήσια έκθεσης και στην περίπτωση της χώρας μου, εφιστώ ε, ε, την προσοχή σας, αλλά όχι μόνο. Επίσης δεν έχει δόντια. Δεν έχει δόντια ε, η Εθνική Αρχή Προστασίας των Δεδομένων σε κάθε χώρα. Στην Πορτογαλία Πρόσφατα ε, ε, επιβεβαίωσε η Εθνική μας Αρχή ότι αυτό που αρνείται η κυβέρνηση, δηλαδή ένα μικρό κατάλογο με ονόματα που ε, VIP λυπούμαστε αλλά θα πρέπει να διακοπεί η διερμηνία γιατί έχει υπάρξει υπέρβαση ήδη του χρόνου. Ευχαριστούμε. It has no clout to make compliance, to demand compliance. And that is even more serious